Right, good morning everybody. Could you take your seats please? Καθίστε παρακαλώ. Και ας ηρεμήσουμε λιγάκι. Right. We will be, will be ready. Μπορούμε να ξεκινήσουμε Καλώς ήρθατε. Σας καλωσορίζω και εγώ και συμπρόεδρος ο κύριος Γιώργη Βιρεγιάννα και σήμερα το πρωί στο πρόγραμμα θα γίνει μια παρουσίαση καταρχάς από τον κύριο Μάριο Τράγκη, τον πρόεδρο ε, του Συμβουλίου για την Οικονομική Σταθερότητα και μετά ο κύριος Ντομινίκ Στρασκάν, ο διευθυντής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου θα μιλήσει και στο τέλος θα γίνει από το Μισελ Μπανιέ τελική παρουσίαση τον Ευρωπαίο, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά και Υπηρεσίες θα πάρει το λόγο. Δεν χρειάζεται όλους αυτούς να σας τους παρουσιάσω και μετά θα συνεχιστεί η συζήτηση με μέλη του πάνελ που θα μείνουν για τη διεξαγωγή της συζήτησης και στις 12 θα τελειώσουμε. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε. Είμαι σίγουρη ότι όπως και χτες θα έρθουν περισσότεροι όσο περνάει η ώρα. Είναι δυναμική όλη η διαδικασία των αφήξεων. Για να έχουμε τον περισσότερο δυνατό χρόνο στη διάθεση των μελών του πάνελ και στη διάθεση των συγκεκριμένων συναδέλφων θα είναι καλύτερα αν δώσω αμέσως το λόγο στον Μάριο Ντράγκη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας είμαι ευγνώμων για την πρόσκληση και αυτό για δύο λόγους. Καταρχάς είναι τιμή για μένα να είμαι εδώ μαζί σας. Δεύτερον, θεσμικής φύσεως ο λόγος. Δεν υπάρχει καλύτερο και πιο ενδεδειγμένος τόπος θεσμικός από αυτόν για να συζητήσουμε τη διαδικασία των ρυθμιστικών μεταρρυθμίσεων. Τελικά, η τοπική αυτοδιοίκηση, η εθνική δίκηση και η τοπική αυτοδιοίκηση είναι αυτοί που έχουν τελευταίο λόγο όσον αφορά τη διαδικασία της μεταρρύθμισης. Δεν θα μακρηγορήσω επί της οικονομικής καταστάσεω, διότι το Μινίκ στο ΣΚΑΝ είναι δίπλα μου και μπορεί πολύ καλύτερα από μένα να αφαιρθεί σε αυτά. Θα ήθελα να πω δύο λόγια όσον αφορά την ανάκαμψη που είναι μικρή, είναι, δεν έχει πολύ μεγάλους ρυθμούς στην Ευρώπη, είναι εύθραυστη παντού, δεν είναι η ίδια παντού παρόλο που η κατάσταση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αφορά τις πιστώσεις ε, είναι δύσκολη και έχουμε τις παραδοσιακές απώλειες που οι οποίες αυξάνονται στο πιστώσεις σε, σε όλα τα κράτη-μέλη, στις ομοθεσίες, εν γέννη οι τράπεζες με μόνο μερικές εξαιρέσεις κινούνται προς επίλυση των χρηματοδοτικών τους ε, προβλημάτων. Βελτιώθηκαν συνθήκες ή χρηματοδοτικές και οι περισσότερες τράπεζες υπήρξαν επιτεχείς όσον αφορά το τελευταίο δεκάμινο, το δεκάμινο όσον αφορά τη συλλογή κεφαλαίων. Είναι ακόμα έφταστη η κατάστασή τους. Οφείλεται αυτό σε ξαφνικές αλλαγές ε, αξιολογήσεων και βαθμολογήσεων και σχετίζεται με την όλη κατάσταση της οικονομικής ανάκαμψης. Τα λέω αυτά διότι αυτό επηρεάζει τις στρατηγικές εξόδου από την κρίση έχουμε δημιουργήσει στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο άνευ προηγουμένου ρευστότητα τα τελευταία, το τελευταίο 1,5 χρόνο, 2 χρόνια και σωστό ήταν αυτό διότι έτσι μπορούσε να αντιμετωπιστεί αυτή η ξαφνική κρίση. Αλλά τώρα που φαίνεται να έχουμε ξεπεράσει οι περισσότερε τράπεζε μάλλον τα χρηματοδοτικά προβλήματα, ήρθε η ώρα να ξεκινήσει η διαδικασία εξόδου. Πρέπει να γίνει αυτό σταδιακά αλλά με σταθερό ρυθμό αν υπάρχουν κάποιε τράπεζε που έχουν ακόμα προβλήματα, τα προβλήματά του θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με ειδικά μέσα. Δεν μπορούν να μιμηθούν και να πιέσουν την νομισματική πολιτική. Θα πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσει εθνικών αρχών με ελάχιστε τράπεζε, ελάχιστε στην Ευρώπη, που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Πριν αναφερθώ στο πρόγραμμα το 2010, πρέπει να πω ότι προχωρήσαμε μαζί ε, και κάναμε πολλά. Και προετοιμάζοντας αυτή τη συνεδρίαση σκεφτόμουν πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι πιστεύω που, στους οποίους οφείλεται η στεναρή προσπάθεια που καταβάλαμε όσον αφορά την μεταρρύθμιση του τομέα σε όλο τον κόσμο. Τα πολλά καταλάβαμε ότι όλοι είμαστε στο ίδιο σκάφος. Είναι ολοκληρωμένο σύστημα και όλοι είμαστε λοιπόν στην ίδια θέση. Και θέλουμε να διατηρήσουμε αυτό, αυτή την ενιαία χρηματοπιστωτική αγορά. Δεύτερον, υπήρξε άριστη ηγεσία από πλευρά των G20 και η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραμάτισε σημαντικότατο ρόλο σε αυτό το πλαίσιο. Οι G20 συμφώνησαν στόχου, καθόρισαν χρονοδιαγράμματα, επιτάχυναν τη διαδικασία και στην επιτάχυνση τη διαδικασία δημιουργήσαν το FSB από το οποίο ζητήθηκε να συντονίσει άλλους εποπτικούς φορείς. Τι το τρόπος, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το FSB συμφώνησαν όσον αφορά τον καταμερισμό των εργασιών για να είναι αποτελεσματικότεροι. Εποπτεία έχει ανατεθεί στο FSB, ε, στο μάλλον ε, υποπτή είναι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η εφαρμογή των μέτρων ανήκει στις εθνικές αρχές. Υπήρξε πάρα πολύ διεθνής διάλογος και συνεργασία άνευ Και αν εξετάσουμε τις λεπτομέρειες της συνεργασίας που προανέφερα, τι βλέπουμε ότι καταρχάς εκ των άνω προς, το, τα κάτω κίνηση και διθετήσεις εφαρμόστηκαν και σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Αυτές οι διευθετήσεις συμπεριλαμβάνουν μεγαλύτερη εποπτεία, μακροοικονομικά μέτρα και προοπτικές για συνετή διαχείριση, μεθόδους για να εφαρμόζεται δράση όσον αφορά τους κινδύνους. Παραδείγματα αυτών είναι το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, το Οικονομικό Συστήμα των Αμερικανών, το σύστημα αγκαίρου προειδοποίησεω του, του Νομισματικού Ταμείου και του FSB και τη δημιουργία αυτού του φορέα του FSB. Άλλο σημείο που πρέπει να προσέξουμε ότι διάφοροι φορεί εξυγχρονίζουν τα ρυθμιστικά του πλαίσια και δομέ για να μπορούν να ανταποκρίνονται καλύτερα στου τιμικούς κινδύνους, να βελτιωθεί ο συντονισμό και να καλυφθούν τυχόν κενά. Τρίτον, τα ρυθμιστικά πλαίσια επεκτάθησαν μέχρι πριν από κάποια χρόνια η περίμετρο αυτή η ρυθμιστική παρακαλείται ο μιλόν να, είναι, να μιλήσει πιο αργά, του λέγουν για τους διερμηνείς, εκείνος λέει θα ήθελα περισσότερο χρόνο, το, εν τη αυτή περίπτωση και συνεχίζει. Τρίτον, έλεγα ότι η ρυθμιστική περίμετρος έπρεπε να αυξηθεί. Πριν από δύο χρόνια θα ήταν αδιανόητο να θεσπιστεί η νομοθεσία όσον αφορά το εμπόριο παραγόγων, τα κεφάλαια κινδύνου, τα hedge funds διάφορα συστήματα τραπεζικά, τους φορείς βαθμολόγηση τραπεζών. Όλα αυτά έγιναν την τελευταία διετία. Τέταρτον, τώρα υπάρχει διασυνοριακή εποπτεία και συστήματα διαχείρισης κινδύνου για τα μεγαλύτερα χρηματοστατικά ιδρύματα. Τέλος, έχουμε εξαλείψει ουσιαστικά τα αντικίνητρα τα αρνητικά κίνητρα τα οποία ήταν στο, στην πηγή της κρίσης, κυρίως όσον αφορά ε, την εξασφάλιση των διαφορών προϊόντων. Δεν θα πρέπει να υποτιμούμε τα επιτευθέντα. Αλλά κάθε ένας από αυτούς τους τομείς είναι α, δύσκολος. Όσον αφορά τη διαμόρφωση πολιτική, σημειώθηκε μεγάλη πρόεδρο. Είναι και, και η ώρα τη εφαρμογή. Και το σημαντικό μήνυμα είναι ότι θέλουμε να κρατήσουμε μια ολοκληρωμένη παγκόσμια χρηματοσυντική αγορά είναι προαπαιτούμενο για τη σταθερότητα και την ανάπτυξη κάτι τέτοιο. Γιατί τα λέω αυτά. Διότι τώρα ήρθε η ώρα υλοποίησης μέτρων. Υπάρχουν πιέσεις, αυτό είναι ξεκάθαρο. Πιέσεις που θέλουν να διαλύσουν τον αυστηρό χαρακτήρα των προτύπων που έχουν θεσπιστεί και την αξιοπιστία τους. Θα ήθελα να αναφερθώ εκτενέστερα σε αυτό τώρα. Φέτος είναι η χρονιά όπου η αναδιάθρωση του πλαισίου ρευστότητας της Βασιλείας θα είναι μια διαργασία που θα ολοκληρωθεί. Υπάρχει ένα πρόγραμμα, χρονοδιάγραμμα που έχει προβλεφθεί. Η Επιτροπή της Βασιλείας σταθμίζει την όλη προσπάθεια τη βαθμολογία αν θέλετε, ελέγχει με τις τράπεζες κατά πόσο τα στοιχεία είναι λογικά και μπορούν να τα δεχτούν οι φορεί οι τραπεζικοί. Θα γίνει μελέτη μακροοικονομικών συνεπειών που θα εξαχθεί από το FSB μαζί με τη Διεθνή Νομισματική Τράπεζα, ε, Διεθνή Νομισματικό Ταμείο, για να δούμε αν αυτή η απορρίθμιση θα είναι επιζήμια ή θα υπονομεύσει την ε, ανάκαμψη. Και τέλος υπάρχει χρόνος για την υλοποίηση τα νέα πρότυπα θα τεθούν σε ισχύ το τέλος του 2012, έτσι προβλέπεται. Και τέλος, εφόσον αυτά τα νέα πρότυπα θα συνεπάγονται ε, πιο ποιοτική κεφαλοποίηση, πιο ποιοτικά κεφάλαια και διαφορετικό, διαφορετικούς ορισμούς του τι θεωρείται κεφάλαιο, θα χρειαστεί μεγαλύτερος χρόνος εποπτείας και εφαρμογής και σταδιακής υλοποίησεως των αλλαγών που θα οδηγήσουν στο νέο ορισμό των κεφαλαίων. Άρα είναι κατανοητό το ότι πολλές τράπεζες, κάποιες τράπεζες, όχι όλες, αντιδρούν. Εκφράζουν ανησυχίες. Θα πρέπει αυτές οι ανησυχίες να ληφθούν υπόψη, σοβαρά, όμως ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να αφήσουμε τις παρούσες δύσκολες συνθήκες να επηρεάσουν την αξιοπιστία των προτύπων αυτών. Θα πρέπει να θυμηθούμε όλοι πώς καταλήξαμε σε αυτή τη διαδικασία. Θα θυμόσαστε στην αρχή της κρίσης τι έγινε. Συμφωνήσαμε όλοι ότι θέλαμε να έχουμε χρηματοστική αγορά και το μέχρι χρηματοστικών υπηρεσιών περισσότερα κεφάλαια, λιγότερο χρέος και να μην υπάρχουν αρνητικά, μάλλον κίνητρα που οδηγούν σε αρνητικά αποτελέσματα. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε τώρα. Ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρχει και παρκής χρόνος μετάβασης, ούτως ώστε να μην ε, επηρεάσουμε αρνητικά την ανάκαμψη. Αυτή είναι η σημαντική ε, διαφορά που πρέπει να έχουμε υπόψη μας και η διάκριση. Τέλος, τέλος, τέλος πάντων. Το άλλο σημείο που αφορά το πρόγραμμα του 2010 είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος του να είναι κάτι πολύ μεγάλο του να αποτύχει ή τα συστημικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και θεσμοί. Για πρωτού αναφερθώ σε αυτό, να σας πω γιατί είναι σημαντικό σαν πρόβλημα. Υπάρχουν θεσμοί, θεσμ, ε, φορείς είναι οι οποίοι πολύ μεγάλοι και αν αποτύχουν θα δημιουργούν συστημικά, συστημικές ζημιές και το κόστος αν καταρρεύσουν αυτοί οι φορείς ε, θα επηρεάσουν όλους μας. Αυτά τα χρηματοδοτικά ιδρύματα γνωρίζουν ότι είναι πάρα πολύ μεγάλα για να αποτύχουν και αναλαμβάνουν περισσότερου κινδύνου γι' αυτό από ό,τι θα ήταν δεδειγμένο. Και γνωρίζουν οι αγορέ ότι αυτά τα ιδρύματα είναι πολύ μεγάλα και τιμολογούν, αποτιμούν αυτούς τους κινδύνους με μία ενδεδειγμένο τρόπο, διότι ξέρουν ότι οι κυβερνήσεις δεν θα αφήσουν αυτά τα τεχνολογικά ιδρύματα να καταρρεύσουν. Γι' αυτό αυτά τα ιδρύματα, ε, ε στα ιδρύματα αυτά κατατίθεται, αν θέλετε, να πολύ μεγάλη κίνδυνη, οι οποίοι αποτιμώνται λανθασμένα και γι' αυτό οι κυβερνήσεις πρέπει να παρέμβουν. Ε, υπάρχουν Τρει διάβλοι παρεμβάσεω κυβερνητικής. Η πρώτη διάβλος είναι η μείωση της πιθανότητας αποτυχίας και κατάρρευση του στικού ιδρύματο και ενδεχόμενη ζημίας που απορρέει από μια τέτοια ζημιά και κατάρρευση. Η γενική στρατηγική του FSB ποια ήταν στον τομέα. Οι εποπτικές αρχές να έχουν τη δυνατότητα, να έχουν την εξουσία να δράσουν ποικιλόμορφα Καμιά φορά υπάρχουν απλουστευμένες δομές, καμιά φορά υπάρχει περισσότερη εποπτή. Άλλες φορές θα υπάρχει ε, υπεβάρυνση όσον αφορά των κεφαλαίων. Δεν υπάρχει μια λύση για τα πάντα. Διαφέρουν οι χώρε, διαφέρουν, ε, διαφέρει η ιστορία στι χώρε αυτέ, διαφέρουν τα χρηματοσυντικά ιδρύματα. Αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτό το πρόβλημα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε όλα τα κράτη-μέλη, σε όλε τι νομοθεσίε. Εδώ μιλάμε για ελάχιστη εναρμόνιση. Με άλλα λόγια, θα έπρεπε να υπάρχει ένα κατώτατο όριο για να αποφύγουμε μείωση κάτω από αυτό το κατώτατο όριο, αλλά κάθε νομοθεσία πέρα από αυτό θα μπορεί να είναι πιο απαιτητική από το κατώτατο όριο. Να θεσπίσει νομοθεσία αυστηρότερη από το κατώτατο όριο. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει το κατώτατο όριο. Και αρκετά μέτρα έχουν συζητηθεί όσον αφορά αυτό και θα προταθούν στην έκθεσή μας η οποία θα υποβληθεί στη Σύνοδο Κορυφής το G20 τον Νοέμβριο. Όμως, Επίσης γνωρίζουμε ότι ανεξάρτητα από αυτό που θα κάνουμε θα έχουμε και αποτυχίες και θα έχουμε καταρρεύσεις και δεν θέλουμε να μην μπορούμε να επιτρέψουμε σε μεγάλες τράπεζες να χρεοκοπήσουν. Πρέπει να μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό. Όταν κάνουν κάποια ασφάλματα βεβαίως. Αλλά θέλουμε επίσης να μπορούμε να χειριστούμε την όλη διαδικασία, να υπάρχει κάποια τάξη. Γι' αυτό χρειάζεται μηχανισμός επιλύσεως των κρίσεων μηχανισμοί που θα μπορούν να εντοπίζουν έγκαιρα τις πιθανότητες χρεοκοπίας, κατάρρευσης, να γίνει σωστός χειρισμός αυτών των χρεοκοπιών, κάτι πολύ περίπλοκο, όπως είδαμε στην περίπτωση των Lehman Brothers, και να υπάρξει και μια μεταβατική περίοδος. Και γι' αυτό η FSB συνεργάζεται με όλα τα κράτη-μέλη, ούτως ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρξουν αυτοί οι μηχανισμοί. Προφανώς για διασυνοριακές τράπεζες και ε, τέτοια ιδρύματα ε, χρειάζονται διαδικασίες συνεργασίας. Εάν καταρρεύσει ένα μεγάλο ίδρυμα θα εμπλακούν πολλές νομοθεσίες και γι' αυτό χρειάζεται ο σωστός συντονισμός. Να πω κάτι εδώ. Εάν δεν καταφέρουμε να επιλύσουμε τα προβλήματα συντονισμού διασυνοριακά, τότε η πιθανότητα οι διάφορες νομοθεσίες να αντιδράσουν λέγοντας ότι μία, ένα ίδρυμα είναι πολύ μεγάλο και πολύ περίπλοκο και γι' αυτό πρέπει να γίνει απλούστερο να εδρεύει σε μία χώρα και να πρέπει να μειωθούν οι διεθνείς διασυνδέσεις ενός ιδρύματος, όλη αυτή η κίνδυνη είναι μεγαλύτερη. Διότι οι εποπτικές αρχές και οι θέλουν τελικά, θέλουν να έχουν τέτοια ιδρύματα τα οποία να μπορούν να αποτύχουν να, να καταρρεύσουν και να χρεοκοπήσουν. Αν αυτό ε, συμβεί, αυτό που προανέφερα, θα χάσουμε όχι μόνο τις ότιμε συνθήκες που πρέπει να επικρατούν, αλλά και η παγκόσμια χρηματοστική, ε, ολοκληρωμένη χρηματοστική αγορά. Τέλος, όσον αφορά αυτό το τομέα του των μεγάλων ιδρυμάτων που είναι πολύ μεγάλα για να καταρρεύσουν, είναι η δουλειά που κάνουμε για να ε, μειωθούν τα προβλήματα εν γέννη. Είδαμε μεγάλη ταχύτητα Είδαμε το πώς διαδόθηκαν τα προβλήματα σε όλο τον κόσμο όταν προέκυψαν. Όταν είδαμε πόσο ισχυροί οι μηχανισμοί είναι τα παράγωγα και οι των παραγόγων. Και πολλή δουλειά έγινε παντού για να αντιμετωπιστεί το εμπόριο των παραγόγων ότι σε κεντρικό επίπεδο. στις απαντήσεις, ερωταπαντήσεις θα αναφέρω σε αυτά εκτενέστερα, αλλά αυτό που λέω είναι το σημαντικότερο κομμάτι των εργασιών μας, διότι ε, θέλουμε να βελτιώσουμε τη διαφάνεια, μεγαλύτερη ορατότητα στις αγορές ε, που δεν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά σήμερα. Και τις επόμενες εβδομάδες θα καθορίσουμε ορισμό ποια παράγωγα θα πρέπει να τυποποιηθούν διοτυποποίηση αυτών των προϊόντων είναι βασική σημασία για να υπάρχει κεντρική αντιμετώπιση του εμπορίου αυτών των προϊόντων. Νομίζω ότι ε, ολοκλήρωσα την παρουσίασή μου. Να πω όμως κάτι ότι τώρα είναι κρίσιμες στιγμές που περνάμε και εξαρτώμεθα κατά πολύ από την υποστήριξή σας για την εφαρμογή αυτών των μέτρων. Ε, το 2010 είναι πιθανότατα ο πιο σημαντικός χρόνος, ούτως ώστε τα σχέδια να μετατραπούν σε δράση. Τα λόγια να γίνουν έργα και νομοθεσία. Αυτά και ευχαριστώ. Thank you very much. Um, Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε αμέσως στην επόμενη παρουσίαση του κυρίου Ντομινίκ Στροσκάν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρα. Χαίρομαι που βρίσκομαι σήμερα εδώ, σε αυτή την πολύ σημαντική συνεδρίαση Ευρωπαίων Κοινοβουλευτικών. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι σε αυτά που μόλις ακούσατε, που από τη... Αυτό βέβαια ίσως σημαίνει ότι χρειάζεται να ακούσετε ξανά κάποια πράγματα, από την άλλη ίσως είναι καλύτερα που τα ξανακούτε. Θα μιλήσω λίγο για το θέμα της ανάκαμψης του χρηματοπιστωτικού τομέα και μετά θα περάσω στις προτεραιότητες που πρέπει να έχουμε για την μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα προκειμένου να περάσουμε σε μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Νομίζω ότι όλοι συνειδητοποιούμε ότι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή πριν από ένα χρόνο, πριν από 18 μήνες φοβόμαστε ότι θα είχαμε μεγάλη ύφεση. Ότι η κατάσταση θα μπορούσε να επιδεινωθεί τραγικά. Αυτό το αποφύγαμε. Δεν αποφύγαμε όμως το κόστος και η κρίση είχε τρομερό κόστος παντού στον κόσμο. Από την άλλη πλευρά η κρίση μας ταπείνωσαν θέλετε όλους γιατί αποκάλυψε διάφορες αδυναμίες, σοβαρές αδυναμίες στο οικονομικό αλλά και το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε ευκαιρία και εμείς και εσείς αλλά και καθήκον να ανασχηματίσουμε τους θεσμούς μας προκειμένου να γίνουν πιο ισχυροί και πιο ανθεκτικοί στις κρίσεις. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν μπορούμε όντως να αξιοποιήσουμε την κρίση. Οφείλω να πω ότι ανησυχώ λίγο. Γιατί ναι μεν τα καλά νέα είναι ότι έχουμε πλέον ανάπτυξη, αλλά Υπήρχαν ε, κάποια πράγματα τα οποία άλλαξαν και είναι όντως αλήθεια ότι κάθε κυβέρνηση έχει τη δική της ατζέντα και είναι λίγο δύσκολο να συνεργαστούν. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το μικρόφωνο του ομιλητή. με συγχωρείτε. Αν λοιπόν θέλουμε να επιτύχουμε συνεργασία προκειμένου να θέσουμε τα θεμέλια για πιο σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη μπορούμε να το κάνουμε. Τι θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν. Καταρχάς, έχει ξεκινήσει η ανάκαμψη και τα πράγματα πάνε καλύτερα από ό,τι περιμένουμε. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει ανάπτυξη 4% παγκοσμίως για το 2010. Όμως μιλάμε για ανάκαμψη πολλών ταχυτήτων αυτή τη στιγμή. Στις πιο προηγμένες οικονομίες είναι πιο μετριασμένα τα πράγματα. Για παράδειγμα, για την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπουμε ανάπτυξη 1% που δεν είναι μεγάλο νούμερο. Επίσης, αν δείτε τα νούμερα ακόμη πιο προσεκτικά, θα δείτε ότι στις αναπτυγμένες οικονομίες έχουμε μικρή ανάκαμψη και η οποία βασίζεται κυρίως στην ενίσχυση από το δημόσιο και στην ιδιωτική ζήτηση και όχι στην ιδιωτική ζήτηση. Άρα δεν είναι εύκολο να ξεπεράσουμε. Αντιθέτως, στις αναδυόμενες οικονομίες έχουμε πολύ πιο ισχυρή ανάπτυξη. Εδώ όμως πρέπει να αναφέρω κάτι. Καλή είναι η ανάκαμψη. Είναι το πρώτο βήμα. Όμως, μετά θα επανέλθουμε στο πρόβλημα που είχαμε πριν από την κρίση. Που αυτή τη στιγμή έχει κρυφτεί πίσω από την κρίση. Και τότε το βασικό ερώτημα θα είναι η ισορροπία της παγκόσμιας ζήτησης. Δεν πρόκειται για νέο θέμα και ήδη έχουν ακουστεί πολλά περί αυτού. Όμως τώρα, μετά την κρίση, οι ηγέτες του G20 το έχουν αναγνωρίσει ως βασική προτεραιότητα. Και ένα από τα καλά πράγματα της κρίσης είναι ότι τώρα πλέον όλοι είναι περισσότερο συνειδητοποιημένοι για το ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις παγκόσμιες ανισορροπίες. Τι εννοούμε σε επίπεδο χωρών. Γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχουν χώρες με τεράστια ελλείμματα, για παράδειγμα οι Ηνωμένε Πολιτείε αλλά και κάποιες ευρωπαϊκές χώρες που πρέπει να αποταμιεύσουν περισσότερα χρήματα και να βασιστούν λιγότερο στην κατανάλωση. Από την άλλη πλευρά έχουμε χώρες με τεράστια πλεονάσματα εμπορικού ισοζυγίου, όπως η Κίνα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Γερμανία και ακόμη και τώρα μπορεί να αυξάνεται η εγχώρια ζήτηση ή να αυξάνονται οι επενδύσεις, αλλά αυτό να γίνεται με διαφορετικό ρυθμό σε κάθε χώρα. Ένα άλλο θέμα βεβαίως είναι το θέμα του συναλλάγματος και της τιμή του που θα έπρεπε να ανατιμηθεί σε κάποιες χώρες. Για παράδειγμα, το Yuan Renminbi στην Κίνα. και ελπίζουμε ότι στα πλαίσια αυτής της διόρθωσης των ανισορροπιών θα πρέπει να υπάρξει ανατίμηση του MBBU. Και δεν εννοούμε ότι το χρειαζόμαστε για να υπάρξει η διόρθωση των ανισορροπιών, αλλά ότι αν αυξηθεί η εγχώρια ζήτηση στην Κίνα, αυτό όντως θα αναγκαστεί να οδηγήσει σε ανατίμηση του νομίσματος. Γιατί τα αναφέρω αυτά, γιατί θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η οικονομική πολιτική των χωρών μετά την κρίση. Και για να έχουμε μια καλή πολιτική, το βασικό θα είναι η συνεργασία. Γνωρίζετε ότι οι G20 αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν ένα νέο πρόγραμμα, το πρόγραμμα από κοινού αξιολόγησης, που είναι ενδιαφέρον πρόγραμμα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα προσφέρει ανάλυση και στήριξη. προκειμένου να μπορούμε να διαπιστώσουμε αν θα υπάρχει αν υπάρχει συνοχή στις προβλέψεις των διαφόρων κρατών. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουν προβλέψεις για τα επόμενα 4-5 χρόνια πολλές χώρες, η Κίνα, η Ιαπωνία, η ΙΠΑ είναι παρόμοιες, είναι συγκρίσιμες. Όχι. Άρα πρέπει να επιτύχουμε μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ αυτών των προβλέψεων. Γιατί ήταν και αυτό ένα, ένας από τους λόγους της κρίσης. Τώρα ας επικεντρωθώ σε κάποια βασικά θέματα για σήμερα, αλλά και στον ρόλο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που αποτελεί βασικό στοιχείο της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής δομής. Να πω ότι γενικά το υπάρχον σύστημα μας έχει εξυπηρετήσει αρκετά κατά τη διάρκεια της κρίσης. Το αμερικανικό δολάριο έπαιξε ρόλο στηρίγματος και νομίζω ότι πριν την κρίση αν είχε μιλήσει κάποιος για μια κρίση η οποία θα είχε ξεκινήσει στη ΣΥΠΑ και θα επεκτηνόταν σε όλο τον κόσμο θα προέβλεπε κατάρρευση του δολαρίου. Αυτό δεν έγινε και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο χρειάστηκε να προσφέρει στήριξη σε αρκετά μέλη του, όμως παραμένει ένα πρόβλημα που είναι η αύξηση των αποθεματικών, κάτι που αυξάνει το, την πίεση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εγώ θεωρώ ότι αν είχαν καλύτερες ασφαλίσεις οι χώρες δεν θα χρειάζονταν τόσο μεγάλα αποθεματικά. Γιατί αυτά τα αποθεματικά τα αυξάνουν επειδή φοβούνται ότι μπορεί θα βρεθούν σε μεγάλη πίεση και να καταλήξουν να ζητήσουν βοήθεια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που όπως όλοι γνωρίζουμε είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Βεβαίως, όταν κάποιος θέλει να έχει μεγάλα αποθηματικά συναλλάγματος, αυτό είναι δύσκολο και βεβαίως ε, θα πρέπει να ανταγωνιστεί στις υπόλοιπες χώρες, γιατί δεν μπορούν όλες οι χώρες να έχουν πλεονάσματα προκειμένου να αυξήνουν τα αποθεματικά. Για να βοηθήσουμε την κατάσταση δημιουργήσαμε μία νέα διαδικασία, τη Flexible Credit Line, σε ευέλικτες πιστώσεις δηλαδή, που χρησιμοποιήθηκαν από δύο χώρες, το Μεξικό, που πριν από λίγες μέρες τον ανέωσε για άλλα για άλλους έξι μήνες, καθώς και από την Κολομβία και την Πολωνία, τρεις χώρες συνολικά. Αυτό το εργαλείο λοιπόν ευέλικτης πίστοσης δεν έχει φτάσει ακόμα την τελική του μορφή και μπορεί σίγουρα να βελτιωθεί, όμως μπορεί να βοηθήσει στο πρόβλημα των αποθεματικών. Και πρέπει να το έχετε υπόψη σας όλοι. Περνάω τώρα στα θέματα του χρηματοπιστωτικού τομέα. Τι μπορούμε να κάνουμε για να αναδιαρθώσουμε τον χρηματοπιστωτικό τομέα ώστε να στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη χωρίς να πληρώνουν τις κρίσεις του τα κράτη και οι φορολογούμενοι όπως έγινε αυτή τη φορά. Σε επίπεδο χωρών νομίζω ότι είναι γνωστές οι προτεραιότητες. Τα ανέφερε και ο Μάριο. Αύξηση της ε, του ελέγχου και αυτό ίσως είναι ακόμη πιο σημαντικό από την αύξηση των ρυθμίσεων γιατί όσο καλή νομοθεσία και αν έχει κανείς αν δεν ελέγχεται η εφαρμογή της δεν βοηθάει σε τίποτα. Μετά, μηχανισμοί επίλυσης κρίσεων. Κάτι που πρέπει να γίνει και ήδη έχει ξεκινήσει να γίνεται. Και Επιπροσθέτως, θα πρέπει να υπάρχουν απαιτήσει για μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση και καλύτερης ποιότητας κεφαλαιοποίηση από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Με απαιτήσει για μεγαλύτερη ευστότητα κτλ. Κάτι που επίσης έχει ξεκινήσει να γίνεται. Πάντως, όταν μιλάμε για χρηματοπιστωτικό τομέα, συνήθως σκεφτόμαστε τον τραπεζικό τομέα όμως υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι του χρηματοπιστητικού τομέα, οι ασφάλειες, όπου η κατάσταση είναι κάπως διαφορετική, όπου σκέφτονται περισσότερο μακροπρόθεσμα, γιατί μιλάμε για αποταμιεύσεις μακροπρόθεσμες πάντα. Και η κατάσταση σε αυτόν τον τομέα των ασφαλιών είναι διαφορετική από αυτών των τραπεζών και πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτές τις διαφορές. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε επιτύχει κάποια πρόοδο και εδώ μπορώ να τονίσω και την συμβολή των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Όμως, όλα αυτά χρειάζονται χρόνο. Στην προηγούμενη κρίση του 30 είχα χρειαστεί 12 χρόνια. Εμείς δεν έχουμε 12 χρόνια στη διάθεσή μας. Έχει αρχίσει το κοινό να ρωτάει τι κάνετε. Άρα αυτή τη στιγμή το ερώτημα είναι η πολιτική σε όλες τις χώρες είναι προετοιμασμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα για την ανάπτυξη. Και όταν μιλάω για πολιτικούς εννοώ και εσάς τους βουλευτές. Είστε διατεθειμένοι να προωθήσετε τις μεταρρυθμίσεις με ταχύτητα, ίσως όχι με την ταχύτητα που επιθυμεί το κοινό, αλλά με ταχύτητα. Γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε αντιμέτωποι με την κοινή γνώμη που διαπιστώνουν ότι υπάρχει κρίση και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε γρήγορα. Και το πρόβλημα είναι ότι τι θα συμβεί αν δεν προχωρήσουμε αρκετά γρήγορα σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό που ήδη βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει να γίνεται. Χώρες να επιλύουν το πρόβλημα σε εθνικό επίπεδο προτείνοντας διαφορετικές μεταρρυθμίσεις με κίνδυνο να έχουμε μη συντονισμένες πολιτικές στρεβλώσεις στο θέμα της ροής κεφαλαίων και μη ρυθμιζόμενη διαιτησία. Arbitrage. Μίλησε και ο Μάριο για τις δυνατότητες επίλυσης κρίσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Έχουν προταθεί διάφορες λύσεις, μεταξύ των οποίων τα Living Wills, διαθήκη εν ζωή και άλλα μέτρα. Πέρα όμως από αυτά τα μέτρα, τα κατασταλτικά, θα μπορούσαμε να δούμε και προληπτικά μέτρα, όπως για παράδειγμα τον περιορισμό του μεγέθους ή της πολυκλοκότητας των χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Όμως, πολύ συχνά αυτά τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή προτείνονται δεν επεκτείνονται πέρα από το εθνικό πλαίσιο. Άρα αυτή τη στιγμή αναμένουμε μεν κάτι σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά έχουν ξεκινήσει και πολλές εθνικές προσεγγίσεις. Και αυτό είναι που κυρίως με ανησυχεί εμένα. Βεβαίως θα μου πείτε, εγώ είμαι επικεφαλής ενός διεθνούς οργανισμού και γι' αυτό ζητάω πολυμερή και όχι εθνική προσέγγιση. Όμως, επαναλαμβάνω, ο κίνδυνος είναι αυτός που ήδη βλέπουμε. Κάποιες κυβερνήσεις θα αρχίσουν να εφαρμόζουν εθνικές λύσεις οι οποίες ενδεχομένως να είναι καλές σε εθνικό επίπεδο, αλλά είναι οι χειρότερες δυνατές λύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Τώρα, για την Ευρώπη, τι έχουμε να πούμε. Σίγουρα υπάρχει καλή πρόοδος, υπάρχει πρόταση για το σύμφωνο σταθερότητα στο διασυνοριακό. Επίσης ε, υπάρχει πρόταση για ένα σύστημα δίκτυο ελεγκτικών αρχών. Όμως, εγώ αυτό που θα ήθελα να κάνω είναι να σας ζητήσω και από εσάς και από το Συμβούλιο να καταλήξετε σε μία συμφωνία όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Γιατί θέματα όπως η διαχείριση των κρίσεων και η επίλυση των κρίσεων, ειδικά για τις διασυνοριακές τράπεζες, όπως είπε και ο Μάριο, είναι κάτι που πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Εγώ αυτό που νομίζω ότι χρειαζόμαστε είναι ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την πρόληψη και την διαχείριση των κρίσεων, καθώς και ένα πλαίσιο για την προστασία. Ένα πλαίσιο που θα περιλαμβάνει μία Ευρωπαϊκή Αρχή Επίλυσης Κρίσεων που θα διαθέτει την εντολή και τα εργαλεία που θα της επιτρέπει να αντιμετωπίζει το πρόβλημα της πτώχευσης συστημικών διασυνοριακών τραπεζών. Θα μου πείτε αυτό είναι πολύ δύσκολο. Ναι, αλλά τεχνικός εφικτό. Χρειάζεται όμως ισχυρή πολιτική βούληση προκειμένου να μπορέσουμε να αντισταθούμε στις εθνικές πιέσεις και να επιτύχουμε κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και ακόμη πιο σημαντικό σε διεθνές επίπεδο. Και κλείνω με δύο σχόλια. Καταρχάς για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σίγουρα πρέπει να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τα όσα γνωρίζουμε και την ανασχόλησή μας με τους εσωτερικούς κινδύνους. Χρειαζόμαστε πιο ποικίλε μορφές και ευέλικτες μορφές εργαλείων. Επίσης χρειαζόμαστε καλύτερη συνεργασία με τη, τα περιφερειακά αποθεματικά ταμεία. Γνωρίζετε ότι υπάρχει η πρωτοβουλία Τζενχουάι στην Ασία. Θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε και με αυτό το αποθεματικό. Επίσης, ένα άλλο θέμα. Έχουμε εμπειρία με τις ευρωπαϊκές χώρες, γιατί έχουμε συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Άρα, το ΔΝΤ μπορεί να συνεργαστεί με περιφερειακούς οργανισμούς. Απλά πρέπει να υπάρξει καλός συντονισμός. Και ένα τελευταίο σημείο αφορά τον χρηματοοικονομικό τομέα. Θα ήθελα να επαναλάβω το βασικό σημείο που ήθελα να αναφέρω σήμερα. Χωρίς διεθνή συνεργασία δεν μπορούμε να επιτύχουμε. Καταρχά χρειαζόμαστε διεθνή συνεργασία μεταξύ οργανισμών. Νομίζω ότι αυτή λειτουργεί καλά. Το επόμενο θέμα είναι η διεθνή συνεργασία μεταξύ κρατών. Νομίζω ότι σε αυτή την χρήση είχαμε ανεπανάληπτη συνεργασία μεταξύ κρατών. Κάτι ιστορικής σημασίας. Είχαμε πραγματικά ασύγκριτη επιτυχία στο θέμα της συνεργασίας μεταξύ κρατών με περίπου όμοια μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης και ίδιες ενισχύσεις. Αυτό δεν είχε συμβεί ποτέ στο παρελθόν. Τώρα λοιπόν που έχουμε ξεπεράσει σχεδόν την κρίση και που ασχολούμαστε με την αναδιάρθρωση του τομέα αυτού, ο κίνδυνος είναι να εξαφανιστεί αυτή η θέληση συνεργασίας. Εδώ λοιπόν θεωρώ ότι τα εθνικά κοινοβούλια και ακόμη περισσότερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση όχι μόνο απλά του να δημιουργήσει καλύτερους μηχανισμούς, αλλά να πιέσει ώστε αυτοί οι μηχανισμοί να εφαρμοστούν σε διεθνές, σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή είναι η πρόκληση σήμερα και για, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να επικεντρωθούμε σε αυτό θυμηθούμε δηλαδή ότι σε μια παγκόσμια κρίση δεν αρκεί μια εθνική ή περιφερειακή λύση, αλλά μόνο μια παγκόσμια λύση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα προχωρήσουμε και θα πάμε στην τελευταία παρουσίαση του Επιτρόπου Μισελ Μπαρνιέ. Πριν το κάνουμε αυτό όμως, να επενθυμίσω κυρίως τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων ότι αν θέλετε να θέσετε ερώτημα, αφού μιλήσει ο Επίτροπος ο κ. Μπαρνιέ, θα μπορείτε να δείχνετε τον ενδιαφέρον σας προς τη γραμματεία εντωμεταξύ για να δούμε ποιος θέλει να μιλήσει και να συλλέξουμε τα ονόματα. Είναι αδύνατο να το κάνουμε εδώ, χωρίς κι άλλα, αν μπορείτε να στείλετε τα σημειωματάκι. Καλωσορίζω λοιπόν τον Επίτροπο Μπάρνιε και του δίνω το λόγο. Μισελ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κυρία Μπούς, κυρία Πρόεδρε, κυρίοι και κυρίες βουλευτές, ευρωβουλευτές και εθνικοί βουλευτές, ζητώ συγγνώμη καταρχάς που κατέφθασα καθυστερημένα και ότι πρέπει να σας εγκαταλείψω. Δεν είναι έλλειψη ευγένειας. Κάθε Τετάρτη πρωί βλέπετε Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεδριάζει μια φορά την εβδομάδα, είναι υποχρεωτική παρουσία μας εκεί Είχα την άδεια του Προέδρου Μπαρόσο να εγκαταλείψω αυτή τη συνεδρία, αλλά θα πρέπει να επιστρέψω. Συζητούμε πολλά από αυτά τα θέματα, βλέπετε. Όμω με τα χαρά να προσφέρω και εγώ τη συνεισφορά μου στη συζήτηση που αποφασίστηκε να διεξαχθεί εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων. Θεωρώ ότι αυτό είναι ευφιέστατο και χρησιμότατο. Σεβόμαστε έτσι το γράμμα και το πνεύμα της συνθήκη τη Αβώνα, διότι μαζί θα πρέπει να νομοθετούμε και να προχωρούμε. Θα ήθελα να ζη... από τον Μάριο Τράγκη να ζητήσω και τον Ντομινίκ Τόσκαν που άκουσα εν μέρη να ζητήσω συγγνώμη από τους δύο ομιλητές που δεν άκουσα όλα όσα είπαν και τους ευχαριστώ για την παρουσία τους εδώ διότι και οι δύο είναι επικεφαλής χρηματοδοτικών φορέων παγκοσμίου εμβελίας και σημασίας και είναι επικεφαλής της παγκόσμιας αυτής ρύθμισης που ανέφερε ο Ντομινίκ Στρόσκαν. Καταρχάς κάποιες σκέψεις αρχικές σχετικά με το χρονικό σημείο που βρισκόμαστε. Βγαίνουμε από την πιο βία κρίση μετά το 1929 που δεν τελείωσε. Ακόμα και αν μπορούμε να ελπίζουμε να φανταστούμε μια διέξοδο από την κρίση και μια νέα ανάπτυξη. Θα βγούμε αυτή την κρίση όπως μπήκαμε. Βεβαίως, σίγουρα, όχι, όχι. Δεν θα βγούμε, δεν πρέπει να βγούμε αυτή την κρίση όπως μπήκαμε σε αυτή την κρίση. Ούτε όσον αφορά την φύση της αναπτύξεως στην οποία ελπίζουμε, που πρέπει να είναι διαφορετική ανάπτυξη, πιο ποιοτική. Και αυτό το νόημα έχει και το πρόγραμμα Ευρώπη 2020 που συζητείται στο Συμβούλιο Υπουργών και στο Κοινοβούλιο. Ανάπτυξη εφιέστερη, πιο πράσινη, πιο δίκαιη πιο ισότιμη. Ούτε όσον αφορά τη φύση της αναπτύξεως που ευχόμεθα και για την οποία πρέπει να κινηθούμε, ούτε όσον αφορά την ίδια την κρίση που θα πρέπει πάση θυσία να βγάλουμε κάποια μαθήματα από αυτή την κρίση. Είναι κάτι αναγκαίο αυτό για να αποφύγουμε και άλλες κρίσεις. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την οποία εκπροσωπώ, θέλει να καταβάλει κάθε προσπάθεια υποβάλλοντας προτάσεις, αυτό είναι ο ρόλος της άλλωστε, και μετά από αυτό αυτοί που έχουν την πολιτική ευθύνη, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, που συμμετέχουν στο G20, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, υπουργοί, τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι συνομοθέτης, θα πρέπει να υπομισθούν τις ευθύνες τους. εκφράστηκε αυτή η πεποίθηση όσον αφορά τα μαθήματα πρέπει να πάρουμε από αυτή την κρίση και αυτή η νέα ανάπτυξη που θα πρέπει να δημιουργήσουμε με οδηγεί σε ένα σχόλιο όσον αφορά το θέμα αυτό. Δεν εξυπηρετεί τίποτα κύριε και, προ... και να ετοιμάζουμε ένα πρόγραμμα το 2020 και να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τα μέσα της εσωτερικής αγοράς. Υπάρχουν πολλά μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα και να θέλουμε να δημιουργήσουμε τη νέα ανάπτυξη. Δεν έχει νόημα όλο αυτό αν πρέπει να αντιμετωπίσουμε νέες χρηματοστηρικές κρίσεις που θα ε, κατέστρεφαν με τη μια όλες τις προσπάθειες. Άρα το πρακτικό θέμα είναι αυτό που έφυξε ο Ντομινίκ Στροσκάν. Να οικοδομήσουμε τη νέα τάξη πραγμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο που η υπάρχει πλαισίωση της μετακίνησης των κεφαλαίων και των κερδοσκοπικών προσπαθειών. Δεν πιστεύω στην αυτορύθμιση αυτού του παγκόσμιου σύστημα. Υπήρξαν αυτοί μάλλον, που πίστευαν στην αυτορύθμιση και εκείνοι που πίστεψαν και αυτό το πράγμα και τελικά αντιμετώπισαν την πραγματικότητα. Έχουμε έναν οδικό χάρτη, ανεξάρτητα τι ευθύνε που έχουμε εθνικέ και ευρωπαϊκέ. Είναι ο οδικό χάρτη των G20 και έχω δεύτερο οδικό χάρτη που αφορά την εφαρμογή των όσων λέει η έκθεση Δελαροζιέρ για την εποπτεία. Θα ξαναρυθμίσουμε το σύστημα, πρέπει να το κάνουμε αυτό με ένα ευφυή τρόπο, βάσει μελετών συνεπειών που θα είναι πολύ ευθυρές. Αυτό σημαίνει κυρίες και κύριοι να ρυθμίσουμε συντονισμένα σε διεθνές επίπεδο. Αυτή είναι η πρόκληση της παγκόσμιας ρύθμισης. Είναι κάτι Προφανέ, οι παγκόσμιε αγορέ χρειάζονται παγκόσμια ρύθμιση. Euh, euh, Χρειάζεται να μην αντιμετωπίσουν θετικά το πρόβλημα, να μην χάνουν όλοι. Χρειάζεται να ρυθμίζουμε αποφεύγοντα τον πειρασμό τη υπερβολικής ρύθμιση. Ο δικό χάρτη λοιπόν των G20 οδηγεί σε κάποιε ε, προσεγγίσεις. Εγώ είμαι αποφασισμένος να ακολουθήσω κάποιες διαδρομές. Πέντε διαδρομές. Πρώτα απ' όλα το θέμα της εποπτείας είναι σημαντικό θέμα. Η εποπτεία των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων είναι ο κρογωνίος λήθος της προσπάθειας ρύθμισης. Αν δεν καταφέρουμε να επιφέρουμε μεταρρύθμιση σε αυτό το τομέα βάσει της εκθέσεως Ντελαροζία δεν θα πετύχουμε τίποτα. Οι αλλαγές που προτείνουμε είναι θεμελιώδου σημασίας πώ να ξαναδημιουργηθεί εμπιστοσύνη στο χρηματοστικό σύστημα αν οι ευρωπαϊκοί κανόνε ερμηνεύονται διαφορετικά στη Μαδρίτη, στο Δουβλίνο. Πώ να εντοπίσουμε του κινδύνου αν δεν εποπτεύουμε σε ευρωπαϊκή κλίμακα τι μακροοικονομικέ μεταβλητέ και την έκθεση σε παγκόσμιο επίπεδο των χρηματοδοτικών φορέων. Πώ θα αντιμετωπίσουμε τι δυσκολίε των χρηματοδοτικών ομήλων εάν δεν υπάρχει κοινοποίηση των πληροφοριών μεταξύ των υποπτικών αρχών και δεν γίνεται αυτό αποτελεσματικά και πώς να είμαστε αξιόπιστοι άλλο σε διεθνές επίπεδο αν οι υποπτικές αρχές, οι εθνικές υποπτικές αρχές δεν συντονίζονται. Δεν υπάρχει μηδέα ανταλλαγή ε, προβληματισμών και δράσεων και εκφράζουν διαφορετικές τοποθετήσεις. Έχουμε φιλόδοξο πρόγραμμα, δεν είναι επαναστατικό. Το ρεαλιστικό μας πρόγραμμα προϋποθέτει μια πολιτική βούληση ισχυρή. Είναι η στιγμή της αλήθειας τώρα και σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, υπουργών που καλούμε να δείξουν πολιτική βούληση και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επίση. Και μετά πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα, κυρίε και κύριοι. Μια αποτυχία θα ήταν σοβαρή για την Ευρώπη. Και κακό μήνυμα, πολύ κακό μήνυμα για την σταθερότητα τη χρηματοπιστωτική. Είπαμε στους συνομιλητές μας, στα κράτη-μέλη, όσον αφορά το θέμα της εποπτείας, το οποίο επεξεργάζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών, που είναι αποφασισμένο το Συμβούλιο Υπουργών, ομόφωνα τα αποφάσει 2 Δεκεμβρίου ότι πρέπει να κινηθούμε και πρέπει να γίνουν παραχωρήσεις και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την προστιθέμενη αξία που δίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και χαιρετίζω εδώ το έργο τη κυρία Μπουλάρ και του κυρίου Γκαρσία Μαργκάλο και του κυρίου Γκιγκόλτ και του κυρίου Σκινέρ που πολλοί από αυτού είναι εδώ και εργάζονται, επεξεργάζονται αυτό το θέμα και αυτή η προστιθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λέγω είναι πάρα πολύ σημαντική. Πιέζει ο χρόνο, λείπει χρόνο. Έχουμε λίγο χρόνο για να ανταποκριθούμε στι δεσμεύσει ανέλαβαν αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων για τη δημιουργία ενό υποπτικού συστήματο και να είναι έτοιμο αρχέ Ιανουαρίου 2011. Δεύτερο, η προσέγγιση, δεύτερο εργοτάξιο είναι του κεφαλαίου των τραπεζών που είναι στο επίκεντρο του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Θα πρέπει να έχουμε περισσότερα κεφάλαια ποιότητα στο τραπεζικό σύστημα και πιο συγκεκριμένα στις επιχειρήσεις ή δραστηριότητε κινδύνου. Ανελήφθησαν και εδώ δεσμεύσει από τους G20 και άλλα κεφάλαια, λιγότερος κίνδυνος, περισσότερη ασφάλεια. Οι προχωρούν οι εργασίες, κυρίως την Επιτροπή της Βασιλείας που κάνει καλή δουλειά, Προσπαθούμε οι τράπεζες να γίνουν ασφαλέστερες και να είναι πιο ανθεκτικές όσον αφορά τις κρίσεις. Ήταν ένα θέμα περιπλοκότατων κεφαλαιόδου σημασίας ήταν να βρούμε σωστή ισορροπία όσον αφορά τα νέα πρότυπα, τι νέε προδιαγραφέ, το είπα τι προάλλες στο Λονδίνο. Πρέπει να βρούμε καλή διπλή στάθμιση. Χρονική, τι διάρκεια χρειαζόμαστε για τι μεταρρυθμίσεις και την εφαρμο... όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων. Και προσπαθώ όχι μόνος μου και θέλω να πετύχω αυτή τη διπλή στάθμιση. Προσέχουμε και τις μελέτες αντικτύπου. Η Σάρα Μπόλς το επαναλαμβάνει αυτό συχνά όσον αφορά τις Ευρωπαϊκές Τράπεζες και είναι αντικείμενο διαβούλευσης αυτό που ξεκίνησε. Τρίτη προσέγγιση, τρίτο εργοτάξιο. Όλα αυτά τα εργοτάξια αποτελούν, είναι αλληλένδετα είναι η ευθύνη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Υπήρχαν κενά, ελλείψεις σοβαρές όσον αφορά το μηχανισμό υποπτια και ρύθμισης. Οι εσωτερικοί μηχανισμοί εντοπισμού των κινδύνων της επιχειρήσης, κυρίως όσον αφορά τις επιχειρήσεις, κατέδειξαν σοβαρά κενά. Σοβαρές ελλείψεις θα έλεγα. Και γι' αυτό λοιπόν επεξεργαζόμαστε αυτό το θέμα της διαχείρισης, της διακυβέρνηση των επιχειρήσεων για τις επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, αλλά όχι μόνο αυτέ, όχι μόνο του χρηματοπιστωτικού τομέα. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, διοικητέ που είναι αρμόδιοι, που είναι ικανοί, που είναι παρόντες, που έχουν τεχνογνωσία, έχουν τα μέσα και το χρόνο να εκπληρώσουν το ρόλο τους και τα καθήκοντά τους. Λέω στελέχη, γιατί στελέχη. Και τον έφερα αυτό και σε ένα νομοθετικό κείμενο. Και γυναίκε βέβαια σε αυτές τις θέσει. Πιο πολλές γυναίκε όσον αφορά τις διευθυντικέ θέσει, Χρειαζόμαστε καλύτερη διαχείριση των κινδύνων. Πολλά μεγάλα χρηματοστατικά ιδρύματα εξαφανίστηκαν διότι δεν τήρησαν του βασικούς κανόνες ελέγχου του κινδύνου και διαχείριση. Χρειαζόμαστε αυξημένη ανάληψη ευθύνη από πλευρά μετόχων όσον αφορά τώρα τι αμοιβέ όσον αφορά τα περίφημα bonus. Και εδώ πρέπει να είμαστε πολύ ξεκάθαροι. Οι αμοιβέ οικονομικές δεν θα πρέπει να οδηγούν σε ανάληψη μεγαλύτερων υπερβολικών κινδύνων όπω ίσχυε κατά το παρελθόν και θα πρέπει να εφαρμόσουμε αυστηρά την αρχή των G20 περισσότερη διαφάνεια, καλύτερος έλεγχος και διαφοροποιημένη αντιμετώπιση. Και θα ήθελα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κυρία Πρόεδρε, να εφητέσει τάχιστα την τρίτη αναθεώρηση της οδηγίας για τον τραπεζικό ε, τομέα. Θα ήθελα να χαιρετήσω τη δουλειά και το σχέδιο εκθέσεως της κυρίας Μακάρθη που θα λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Και μετά θα ήθελα να μιλήσω για άλλα θέματα πέρα του χρηματιστικού τομέα, αναφερόμενο στην αμοιβή των εισηγμένων εταιριών, των στελεχών των εισηγμένων εταιριών. Χρειάζεται να υπάρξει κάποια αντιστάθμιση βέβαια τη επίδοση. Και θα πρέπει και να επιβάλλονται κυρώσει σε περίπτωση αποτυχία ανάλογα. Τρίτος, τέταρτο εργοτάξιο μάλλον, που αναφέρεται συχνά τι τελευταίε ημέρε, είναι το σχέδιο οδηγίας που υπευλήθη σχεδόν πριν από ένα χρόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έκανε τη δουλειά της εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τη ρύθμιση των hedge funds και του τομέα του private equity. Ο Πολ Γκοζές έχει κάνει δουλειά πάνω στο θέμα. Μιλάμε για ένα τομέα που παρόλο που δεν παίζει ρόλο στην κρίση αλλά κάποια μέρα είδα ε, ότι αφορά πάνω από το ίμιση των συναλλαγών στο χρηματοδοτικό τομέα. Το private equity και τα hedge funds. Οπότε υπάρχει κίνδυνος συστημικής φύσεως που ε, διέπει αυτό το τομέα. Γι' αυτό προτείναμε πάνω από ένα χρόνο, εδώ και πάνω από ένα χρόνο, μια πρόταση για υποπτία του τομέα αυτό σύμφωνα με τις δεσμεύσεις και τον οδικό χάρτη των G20. Έχουμε τρεις στόχους που έχουμε θέσει. Ενίσχυση της εποπτείας των συστημικών κινδύνων, κάτι που ανέφερα, βελτίωση της προστασίας των επενδυτών και τη δημιουργία εσωτερικής αγοράς για τους χειριστές εναλλακτικών ταμείων και πόρων. Αυτό δεν είναι και το πιο εύκολο. Επ' αυτού το Συμβούλιο των Υπουργών επί Ισπανικής Προεδρίας αποφάσισε χθε να δώσει κι άλλο χρόνο, θα εκφράσω μπροστά σας μία επιθυμία, μία ευχή αυτός ο χρόνος να χρησιμοποιηθεί σωστά για την επίτευξη μιας καλής συμφωνίας λαμβάνοντας υπόψη την αρχική πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη τις εργασίες που διεξήχθησαν υπό την ηγεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να καταλήξουμε σε μια εποπτεία και σε μια ρύθμιση ευφυή και αποτελεσματική του τομέα. Αλλά και εκεί έρχεται η στιγμή της αλήθειας όσον αφορά την αποφασιστικό των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεως για να εφαρμόσουν αυτό το κομμάτι, αυτό το, αυτή τη λίθα, αυτό το τούβλο, αν θέλετε, στο οικοδόμημα των G20. Και κάτι τελευταίο, τελευταίο σημαντικό εργοτάξιο που δεν θέλω να αναφέρω και εδώ έχω να υποβάλω σχετική πρόταση όσον αφορά ένα δομικό πακέτο μεταρρυθμίσεων. Ε, μήνα Ιούνιο θα γίνει αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άνευ καθυστερήσεων θα κάνει τη δουλειά της. Αναφέρομαι στο χατοφυλάκιο των παραγόγων προϊόντων. Εξάλλου είχα συνομιλίες πρόσφατα αυτή την εβδομάδα με τον κύριο Γκένσλερ, τον πρόεδρο της CFTC, της ΕΠΑ, που και εκείνος Προχωράμε σε αυτή την κατεύθυνση, την εποπτεία, τον έλεγχο των παραγόγων προϊόντων. Κάτι σημαντικό. 600.000 ε, δισεκατομμύρια δολάρια εκπροσωπεί. 80% αυτών των παραγόγων διαφεύγουν ελέγχου, διαφανείας, τυποποίησης ή καταχώρησης. 80% θα πρέπει να κινηθούμε στην άλλη κατεύθυνση, να αντιστρέψουμε αυτή την αναλογία, αυτό το ποσοστό στην άλλη κατεύθυνση είναι η κοινή αποφασιστικότητα αυτή που εκφράζω. Μα όπως και ο αρμόδιος για την εποπτεία ο Αμερικανός. Και γι' αυτό θα υποβάλει επί τραπέζης κυβερνήσεων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Κοινοβουλίου σχετική πρόταση τον μήνα Ιούνιο. Θα προτείνω λίγο αργότερα, λαμβάνοντας ε, διαθέτω στον χρόνο να παρατηρήσω, να δω τι κάνει ποιο, κάνει τι μάλλον, χωρί να υπάρχουν αυτοσχεδιασμοί. Θα προτείνω, λέγω αργότερα, ένα κείμενο για να πλαισιωθεί και η κερδοσκοπία. Κυρίω όσον αφορά όταν υπονομεύει τα swaps. Αυτά είναι τα εργοτάξια επί των οποίων κινείται ως είναι καθήκον της άλλωστε Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να καταφέρει, τα καταφέρει όλα μόνη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειάζεται την αποφασιστικότητα, όπω είπα και επαναλαμβάνω, των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των G20, των Υπουργών Οικονομή Οικονομικών, Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων. Χρειάζεται υποφασιστικότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ξέρω ότι δεν λείπει αυτή η υποφασιστικότητα. Χρειάζεται υποστήριξη των Κοινοβουλίων των Εθνικών επίση. Θα ήθελα να κλείσω υποστηρίζοντα την έκκληση για την προσπάθεια αυτή την παγκόσμια που ανέφερε ο, ο του Διεθνού Ομοσπονδιακού Ταμείου ότι χρειάζεται γενική παγκόσμια ρύθμιση, αλλά μέσα σε αυτά τα πλαίσια η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει εφαρμόσει οικονομική και χρηματοστική διακυβέρνηση, ακόμα και αν αυτή μπορεί να βελτιωθεί, θα πρέπει να λάβει τη θέση τη. Και αυτή η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντική, χωρί να φοβάται. Καμιά φορά να προχωράει να μένει πίσω ή να δίνει το παράδειγμα. Ε, αυτό το πνεύμα μας, να ηγούμεθα τελευταία σκέψη είναι μια, έχει πολιτική χρειά. Κυρίες και κύριοι, βλέπουμε πολύ καλά τις συνέπειες, το τίμημα που πληρώσαμε όσον αφορά την κρίση σε επίπεδο προπολογισμού, τα τι γίνεται με τα χρήματα του φορολογουμένου, υπάρχουν οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες. Δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον παρόμοια τέτοια κρίση. Ακόμα και αν υπάρχει πιθανότητα να υπάρξουν και άλλες κρίσεις. Εμεί θέλουμε να κινηθούμε όσον αφορά την πρόληψη διαχείριση μελλοντικών κρίσεων. Άλλο εργοτάξιο αυτό θα το αναφέρουμε στο μέλλον αυτό. Έχουμε καθήκον, θα έλεγα, έναντι των πολιτών μα και έναντι των φορολογωμένων. Να συναγάγουμε μαθήματα από την παρούσα κρίση και να το κάνουμε γρήγορα. Αν δεν το κάνουμε αυτό, όχι μόνο οι συνέπειε, οι δημοσιονομικέ και οικονομικέ θα είναι καταστροφικέ, αλλά οι συνέπειε, οι πολιτικέ θα είναι καταστροφικέ. Και βλέπουμε εδώ και εκεί στην Ευρώπη κάποια σήματα, σημάδια επιστροφής εθνικών αντιδράσεων, επιστροφή σε προστατευτικές αντιδράσεις, καμιά φορά επιστροφή σε εθνικιστικές και λεκιστικές αντιδράσεις. Πρώτο θύμα μια κρίσεω, της νέας κρίσεω που δεν ε, αντιμετωπίστηκε σωστά πολιτικά, θα είναι η νέα αγορά και είμαι υπεύθυνο για την νέα αγορά ως επίτροπος. Αυτή την έκκληση θα αναπευθύνω να υπάρξει πολιτική αποφασιστικότητα για να εφαρμοστεί ο δικός μας χάρτης και να καταλήξουμε σε ευφυή διαχείριση, αποτελεσματική εποπτεία, που αυτό είναι το μήνυμα της οικονομικής κρίσεως από την οποία θα πρέπει να βγούμε. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank Σας ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα θα προχωρήσουμε στις ε, δηλώσεις, σχόλια, ερωτήσεις ε, σε, αυτό το, σε αυτή τη φάση της συνάντησής μας. Ζητώ από τους βουλευτές να είναι το δυνατόν συντομότεροι, διότι αν πάρετε πολύ χρόνο ερωτώντας κάτι δεν θα υπάρξει χρόνος για απάντηση. Θα πάρουμε ομαδοποιημένα κάποια σχόλια ή ερωτήσεις από κοινού, ομού, από τους εθνικούς βουλευτές και τους ευρωβουλευτές προτού τοποθετηθούν οι εισηγητές στο πάνελ. Λυπούμε, λυπούμε που δεν μπορούμε ένα προς ένα να πάρουμε τις ερωτήσεις, αλλά πρέπει να γίνει ομαδοποιημένα. Από τα εθνικά κοινοβούλια. Ο πρώτος είναι ο κύριος Ραλφ Μπρίνκ, νομίζω λέει, από τη Γερμανία. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ θερμά για την ποιοτικά εξαιρετική παρουσίαση στις παρεμβάσεις, στις εισηγήσεις. Ήταν εξαιρετική και μας βοήθησε πολύ. Τρεις ερωτήσεις έχω. Πρώτον, θα ήθελα να πω ότι βλέπουμε όλοι την μεγάλη σημασία του Risk Board. Πώς θα καταφέρουμε τα πορίσματα αυτού του Risk Board σε εθνική δράση να τα υλοποιήσουμε. Πρώτον, την δράση εποπτικών εθνικών αρχών και δεύτερον την δράση διεθνών θεσμικών χρηματοοικονομικών ε, δημοσιονομικών ιδρυμάτων. Η δεύτερη ερώτηση προς τον κύριο Στροσκάν. Εντυπωσιακά παρατηρήσατε και σχεδιάσατε το πεδίο έντασης μεταξύ της ανάγκης για ταχύε λύσει ε, σε εθνικό επίπεδο επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο. Είμαστε αισιόδοξοι και ο κύριος Μπανιέση θα το δει πιστεύω ότι μια καλή ευρωπαϊκή απάντηση ως λύση θα εκπονηθεί. Αυτό όμως δεν βοηθάει αν δεν υπάρξει συμφωνία με τις ΗΠΑ, διότι στο τέλος τέλος θα υπάρχει ε, θέμα διευθέτησης, αρμπιτράζ ε, και οι μεγάλοι οίκοι και τα μεγάλα θεσμικά όργανα μπορεί να ε, έχουν βλαπτικές επιπτώσεις. Πώς θα καταφέρετε να υπάρξει πραγματικά μια λύση, τουλάχιστον με τις ΗΠΑ. Δεν τολμώ να ρωτήσω αν θα υπάρξει λύση με τους Ρώσους ή με τους Ασιάτες όσον αφορά τα δημοσιονομικά. Και η τρίτη ερώτηση, κύριε Στρόσκαν, αν σας, σωστά σας κατάλαβα, σκιαγραφίσατε και είπατε ότι ο ρόλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο risk monitoring βρίσκεται, στην εποπτεία κινδύνων. Αυτό σημαίνει ότι βλέπετε να έχετε κάποιο ρόλο ως International Systemic Risk Board. Ευχαριστώ. I think repeat the first part. Ε- παρακαλώ το πρώτο τμήμα. Το πρώτο τμήμα της ερώτησης ήταν ότι όλοι βλέπουμε τη μεγάλη σημασία του risk board. Πώς θα καταφέρουμε τα συμπεράσματα, τα πορίσματα που θα πορεύσουν σε εθνική δράση στα, στα, ε, στις υπηρεσίες εποπτείας ε, και στα δημοσιονομικά θεσμικά όργανα να υλοποιηθούν. Πώς θα καταφέρουμε αφού θα έχουμε εντοπίσει κίνδυνο να αναλάβουμε δράση. Ευχαριστώ. Thank uh, Σας ευχαριστώ. Επόμενη η κυρία Ελίζα Φερέρα, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ μιλώ υπό την ιδιότητα ως εισηγήτρια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αντιμετώπιση της κρίσης στις διασυνοριακές ε, τραπεζικές συναλλαγές. Γι' αυτό οι παρεμβάσεις που έγιναν εδώ ήταν πολύ σημαντικές για μένα. Θα ήθελα να έχω την άποψή σας για τέσσερα σημεία πολύ εξειδικευμένα, πολύ συγκεκριμένα. Πρώτον, διαρωτώ με, ποια είναι η άποψη ιδιαίτερα του Μάριο Αντράγκη και του κυρίου Στροσκάν. Ποια είναι η άποψή τους για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Παρέμβασης, Ευρωπαϊκού Ταμείου Επίλυσης, Αντιμετώπισης Καταστάσεων Κρίσης στις τράπεζες που θα χρηματοδοτείται από την ίδια, τις ίδιες επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες. Να αποφύγουμε οι φορολογούμενοι να είναι οι τελευταίοι που θα πρέπει να υπομισθούν τα έξοδα αυτά για την λειτουργία αυτό. Έχω συνειδητοποιήσει ότι δεν κάνουμε λόγο για την ε, διάσωση των τραπεζών, αλλά για να υπάρξει δυνατότητα, ας το πω έτσι, περιθωρίου ελιγμών. Από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα ήθελα να ακούσω ποια είναι η άποψή σας για την αρχή αυτή και το ταμείο αυτό. Είναι αναγκαίες, είναι αναγκαία ή όχι. Δεύτερον, η διαδικασία εναρμονισμού μεταξύ πρακτικών δεν θα επιτρέψει μέσα σε ένα λογικό χρονικό διάστημα να υπάρξει εναρμονισμός των δικαίων ε, της νομοθεσίας ε, των κρατών μελών όσον αφορά αυτά τα θέματα. Όταν γίνονται παρεμβάσεις προληπτικές από πλευράς τραπεζών κυρίως, και όταν γίνεται χρήση κάποιων triggers, ε, κάποιων κατοφλίων ή κάποιων μηχανισμών μπορεί να υπάρξει σύγκρουση μεταξύ των δικαιωμάτων των ε, ε, τραπεζών και των μεριδιούχων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Τι θα γίνει λοιπόν για να αποφύγουμε μια κρίση και σε σχέση με το καθεστώς αυτό υπάρχουν συστημικές μεγάλες τράπεζες, υπάρχουν κίνδυνοι συστημικοί για μεγάλες τράπεζες. Πώς το ε, κρίνεται αυτό. Η τρίτη ερώτηση αφορά το συντονισμό. Συντονισμό μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΠΑ. Ξέρω ότι έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια σύγκλησης, αλλά συνεχίζουμε να κατηγορούμεθα ότι προωθούμε, λέει, ρυθμιστικά διαφορετικά συστήματα στη μία όχθη και στην άλλη όχθη του Ατλαντικού πράγμα το οποίο μπορεί να προκαλέσει ε, σύγκρουση αρμοδιοτήτων, ε, ανάγκη διευθέτησης, ε, απώλεια ανταγωνισμού, προβλήματα. Ποιες προσδοκίες υπάρχουν για αυτά τα θέματα. Τελευταία παρατήρηση συναλλαγές και η χρηματοοικονομική αναλογία ευρώ-δολαρίου και ποιες είναι οι προοπτικές σε σχέση με αυτό. Uh, uh, Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκούντερ Στούμπολ από την Αυστρία παρακαλώ επόμενος. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και για τις τρεις εισηγήσει. Ήταν εξαιρετικές και μπορούν να μας βοηθήσουν πάρα πολύ. Στον κύριο Ντράγκη, είμαι ευγνώμων που σε σχέση με τη Βασιλεία 3, τη συμφωνία αυτή, εξέφρασε και κάποιες ανησυχίες. Νομίζω πρέπει να αποφασίσουμε τι είναι αυτό που θέλουμε από τις τράπεζες. Θέλουμε αφενός να διασφαλίσουν, να δίνουν περισσότερες πιστώσεις και δάνεια. Θέλουμε περισσότερο ίδιο κεφάλαιο να δημιουργούν για την αντιμετώπιση της κρίσης. Τώρα κάποιες χώρες αρχίζουν να επιβαρύνουν τράπεζες με ειδικά τέλη και φόρους. Σημερίζομαι εδώ κάπως την ανησυχία του κυρίου Στροσκάν. Όσο βραδύτερα επιτυγχάνουμε πρόοδο, τόσο ταχύτερα θα λαμβάνονται μη συντονισμένα μέτρα από τις χώρες. Και γι' αυτό παρότι είναι πολύ δύσκολο να ε, είχαμε ένα φόρο ή τέλος συναλλαγών θα πρέπει όμως να μην έχουμε στο τέλος τέλος ε, τέλη ή ε, φόρους βάρος των τραπεζών. Πώς βλέπετε τώρα την εξέλιξη και η Αυστρία νίκη δυστυχώς σε αυτές τις χώρες πρέπει να πω που ειδικού φόρους εισπράττουν ή επιβαρύνουν τις τράπεζες με αυτούς διότι αυτό θα ήθελα να αποσαφινιστεί. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ ο Ούντο Μπούλμαν μετά στη συνέχεια και μετά θα επιστρέψουμε να απαντήσουν οι συγητές. Ο κύριος Μπούλμαν. Βλέπω ότι οι κύριοι που βρίσκονται εδώ εμπρός και στην δική μου γλώσσα μπορώ να συνεχίσω ή έχω κι εγώ μια ερώτηση στοχεύει στον πυρήνα των ανησυχιών μου, μια και ο Γερμανός συνάδελφος το προανέφερε αυτό το θέμα πιο πριν. Εμείς βρισκόμαστε μέσα στη μέση μιας φιλόδοξης νομοθετικής προσπάθειας ρύθμισης των πραγμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, επίσης. με την ανησυχία του Επιτρόπου Μπαρνιέ όταν περιγράφει το ευρώ στην εμβέλεια αυτής της κρίση. Για μένα είναι ζήτημα, είναι θέμα αν αυτή η κρίση επιτρέπει καν ακόμα πολιτική λήψη απόφασης για τα οικονομικά θέματα θα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ή θα σηκώσουμε ψηλά τα χέρια και θα παραδοθούμε. Είναι σημαντικό αυτό το θέμα, αν πιστεύει κανείς στη δημοκρατική διακυβέρνηση και διαχείριση. Εγώ το κάνω αυτό και το πιστεύω. Τότε πρέπει να βρούμε όμως πιστικές απαντήσεις και αποτελεσματικές απαντήσεις και στην Ευρώπη και στη ΣΥΠΑ. Για συναδέλφους τώρα από τη ΣΥΠΑ για το ότι υπάρχει η προειδοποίηση ότι κάνουν φιλόδοξες ρυθμίσεις για τα hedge funds και το πώς θα πρέπει να δοθεί συνέχεια με τις καλές βέλτιστες πρακτικές στα χρηματιστήρια επειδή τους λένε δεν πρέπει να υπάρχουν ανταγωνιστικά μειονεκτήματα έναντι της, ε, των Ευρωπαίων. Αν πάμε στους Ευρωπαίους το ίδιο ακούμε αλλά αντίστροφα. Δεν πρέπει λέει, να υπάρχουν μειονεκτήματα για τον ανταγωνισμό έναντι το, α, τους Αμερικανούς. Εδώ υπάρχει ασυμμετρία πίεση σε σχέση με την πολιτική. Εδώ έχουμε ε, διαρκώς συμπίεση καλών προτάσεων επειδή υπάρχει μια σπυροειδή στάση προς τα κάτω υποβάθμισης ή μείωσης επίπεδου. Σας ερωτώ υπό την ιδιότητα key players που έχετε κύριων εμπλεκόμενων στις ε, παγκόσμιες αγορές αλλά και ως ε, εξαιρετικούς γνώστες του σκηνικού της κατάστασης τι μπορούμε να κάνουμε ρωτώ, από κοινού ώστε τα καθεστώτα που πρέπει να βρούμε να είναι δημοκρατικά και υπεύθυνα για τη διαμόρφωση των αγορών και στη ΣΥΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καλύτερα να συντονιστούν μεταξύ τους ώστε η δημοκρατική διακυβέρνηση και η δημοκρατική διαμόρφωση κανονισμών, κανόνων και ε, καταστάσεων να μπορεί να έχει ευκαιρία να επιβιώσει. Ευχαριστώ. Um, do you wish to go first, Mr. Draghi? Ο κύριος Draghi παρακαλώ. Uh, <clears throat> thank you. Thank Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να στραφώ στην πρώτη ερώτηση Νομίζω μπορώ να αναδιατυπώσω με άλλα λόγια. Ποιες είναι η, ποια είναι η προβλεπτή αποτελεσματικότητα αυτού του risk board σε σχέση με την Ευρώπη. Λοιπόν, έχουμε υπόψη ότι θα υποβάλει συντα, ε, συστάσεις ε, το risk board. Κάποιες από αυτές τις συστάσεις θα μπορούν να δημοσιοποιούνται. Αυτό είχαμε πει. Έχουμε υπόψη ότι θα είναι ένα όργανο όπου θα έχουμε εποπτεία σε ανώτατο επίπεδο από ε, ομολόγους και θα μπορεί να ασκηθεί και κάποια πίεση. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω, γιατί στο τέλος τέλος, στη συνέχεια, με τον καιρό που θα περάσει, θα είναι ένα πολύ αποτελεσματικό σώμα ως φορέας, ως όργανο. Μπορώ να μιλήσω νομίζω με την δική μου, με βάση τη δική μου πείρα στην FSB. Η FSB, το έλεγα πιο πριν, σχεδιάζει κανόνες Υπάρχει μια ε, ε, εποπτεία και κάποια πίεση ομολόγων, αλλά είναι όμως ε, θέμα εποπτείας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και θέμα εφαρμογής το θέμα των εθνικών αρχών στη συνέχεια. Τώρα λένε ότι, γιατί λένε ότι ήταν επιτυχής η δράση της FSB και δεν είναι δική μου τοποθέτηση, γιατί το λένε αυτό. Αυτό αφορά την σύνθεσή του για την Ευρώπη στο Risk Board θα έχουμε παρόμοια σύνθεση πάνω κάτω, σαν αυτή που, θα έχουμε, που έχουμε στην FSB. Όχι ακριβώ την ίδια, πανομοιότυπη, αλλά θα συμμετέχουν άτομα που θα συζητούν και θα εξετάζουν τους κανονισμού, αλλά θα υπάρχει και η ευθύνη στην συνέχεια εφαρμογή και υλοποίηση. Είναι η ταυτοποίηση των δύο αυτών ιδιωτήτων στα άτομα αυτά, στου ομολόγου, που δίνει και θα δίνει ισχύ και εξουσία σε αυτό το σώμα και στα μέλη του, στο Risk Board στην Ευρώπη ουσιαστικά θα έλεγα ευελπιστώ και ε, έχω εμπιστοσύνη ότι θα έχει αποτελεσματικότητα αυτή η προσπάθεια πέρα από τα όσα έχουμε σχεδιάσει θεωρητικά. Στην πρακτική εφαρμογή θα είναι πιο αποτελεσματικά. Τώρα, για την παρατήρηση συντονιστικής δράσης με τις ίπα συντονισμού με ίπα υπάρχει μια γενική παρατήρηση και μια συγκεκριμένη, πιο εξειδικευμένη. Ή το γενικότερο σχόλιο είναι δεν νομίζω ότι θα πρέπει να υπερεκτιμούμε ή να τονίζουμε ιδιαίτερα αυτή την έλλειψη ή ενδυνάμει απουσία συντονισμού. Και αυτό αφορά την ερώτησή σας επίσης ε, κατά κάποιο ε, μέτρο. Για δύο λόγους αυτό. Ένας είναι κάποιες από τις προτάσεις ε, που απέρευσαν από τη συζήτηση στη ΣΥΠΑ τους τελευταίους μήνες ήταν ουσιαστικά μέρος, τμήμα των συζητήσεων μέσα στο ίδιο το FSB. Όταν λέω ότι δεν υπάρχει ένα, μια χρυσή ράβδος, μια χρυσή λύση που θα είναι <clears throat> εξίσου καλή για όλες τις νομοθεσίες και περιπτώσεις για παράδειγμα το πρόβλημα χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που είναι υπερβολικά μεγάλα για να επιτραπεί να αποτύχουν και να χρεοκοπήσουν. Εντάξει, υπάρχουν νομοθεσίες όπως τις είπα όπου πιθανόν πιστεύουν ότι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί το θέμα υπερβολικά μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για να αποτύχουν είναι να υπάρξει νομοθετικός διαχωρισμός μεταξύ των trading business και banking business Άλλε όμω ε, χώρε και νομοθεσίε θεωρούν ότι ο καλύτερο τρόπο ε, για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματο θα ήταν διαφορετικέ απαιτήσει όσον αφορά τα ίδια κεφάλαια για το trading και το banking. Και αυτό ήδη βρίσκεται υπόψη στην μεταρρύθμιση τη Βασιλεία 2. Έχει προταθεί και εξετάζεται τώρα σε σχέση με τι αγορέ ακριβώ αυτό βλέπετε ότι οι δύο ε, τα δύο σημεία δεν παρεκκλίνουν τόσο σημαντικά στους στόχους τους. Μπορεί να είναι διαφορετική η χρήση εργαλείων ή μέσων για την επίτευξη του τελικού στόχου. Αλλά αυτό είναι ένα, ένα πεδίο όπου δεν θα έπρεπε να αναμένουμε να υπάρχουν παντού πανομοιότυποι κανόνε ταυτόσιμοι. Υπάρχει όμω ένα τομέα που πρέπει να υπάρχουν πανομοιότυποι κανόνε παντού. Είναι οι απαιτήσει κεφαλαίων και οι απαιτήσει ρευστότητα. Αυτή είναι αυτό που αποκαλώ εγώ μέγιστη, μέγιστος ω πεδίο. Και εδώ για την τελευταία σα ερώτηση κύριε Μπούλμαν. Υπάρχει ένα άλλο πεδίο που πρέπει να έχουμε μέγιστο εναρμονισμό για να είμαστε αποτελεσματικοί. Ο τομέας των παραγόγων. Πρέπει να έχουμε πλήρως εναρμονισμένες πλατφόρμες για αυτές τις συναλλαγές παγκόσμια. Διαφορετικά το regulatory arbitrage θα είναι ακαριέο και αυτό το οποίο εμείς ε, ουσιαστικά ε, θα, ε, αν δεν το κάνουμε, εκεί που θα καταλήξουμε είναι ότι θα πάνε όλα στράφη. Να στραφώ στην τελευταία παρατήρηση European Resolution Fund. Είναι απόλυτα σαφές. Είναι πολύ σαφές ότι όποιους μηχανισμούς θα είχαμε για διευθέτηση προς λειτουργία θα έπρεπε να μπορούν να χρηματοδοτήσουν, να αντιμετωπίσουν την κρίση στη διαχείριση τραπεζικών ιδρυμάτων κατά την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Γιατί ξέρετε, κάποιοι εξαφανίζονται ξαφνικά όταν είναι οφειλέτες και κανείς δεν θέλει μετά να πληρώσει τα σπασμένα. Λοιπόν, στην Ευρώπη όπου αυτά τα ταμεία μικρότερων βέβαια διαστάσεων χρηματοδοτούντουσαν παραδοσιακά από την τραπεζική βιομηχανία. Δεν αποβαίνει τίποτα εναντίον του να χρηματοδοτεί η ίδια η βιομηχανία, η ίδια αυτή η τραπεζική δράση αυτές τις πρωτοβουλίες κατά το τελευταίο 1,5 χρόνο θέλουμε να, χρημα... να επιβαρύνουμε τις τράπεζες με φόρους, τέλη, θέλουμε να εισπράξουμε έσοδα, πολλά τέτοια συναφή. Πρέπει να θυμόμαστε όμως εν τέλει ότι το ίδιο ταμείο είναι εκείνο κεφαλαιακά που θα πληρώνει για όλα αυτά. Θα υπάρξει κάποια στιγμή όπου εξετάζοντας τις επιπτώσεις όλων αυτών των κανονισμών και ρυθμίσεων θα πρέπει να δούμε αυτό θα είναι εφικτό και κάτι άλλο δεν θα είναι. Τι θα είναι το πιο αποτελεσματικό. Δηλαδή δεν αρνούμε, δεν είμαι εναντίον μια τέτοια πρωτοβουλία. Ίσως μπορεί να είναι καλή γιατί μπορεί να είναι κάποιο κίνητρο αυτό, να είμαστε αποτελεσματικοί. Πρέπει όμω να θυμόμαστε ότι η δημοσιονομική συμβατότητα για το σύνολο του τραπεζικού τομέα είναι η λιδία Είναι δύσκολο να εναρμονιστούν οι νομοθετικέ διαδικασίε όσον αφορά τι διαφορετικέ χώρε και τι νομοθεσίε του. Δεν ξέρω αν τα παλαιότερα κράτη-μέλη τη Ένωση έχουν τελείω διαφορετικού νόμου για την αντιμετώπιση χρεοκοπή οποίας ε, μπορεί όμως ε, να ε, πέσω έξω αν εικάσω κάτι. Όμως παρόλα αυτά εκείνο το οποίο πρέπει να εναρμονιστεί και ίσως είμαι κάπως υπερβολικά αισιόδοξο εδώ, αλλά νομίζω ότι έχω δίκιο σε αυτό. Αυτό που πρέπει να εναρμονίσουμε εδώ δεν είναι το σύνολο της νομοθεσίας ε, για τις τράπεζες που έχει ιστορία, προϊστορία 200-300 ετών. Κάτι τέτοιο θα ήταν δυσχερέστατο εγχείρημα. Πρέπει να εναρμονίσουμε μόνο μικρούς τομείς, τομεακά, στις ε, τραπεζικές αυτές δραστηριότητες. Για παράδειγμα, την αντιμετώπιση των collaterals, το ring fencing collaterals, που είναι διαφορετικές διαδικασίες, διεργασίες σε σχέση με τις διαφορετικές χώρες. Είναι σαφώς προσδιορισμένο πρόβλημα περιορισμένων διαστάσεων τομιακά που μπορούμε να το διευθετήσουμε. Αν δεν το κάνουμε αυτό και αν δεν το ρυθμίσουμε γοργά, γρήγορα, και εδώ επανέρχομαι στην παρατήρηση του Ντομινίκ Στρόσκαν η πίεση για την απλούστευση τέτοιων νομικών διατάξεων, η πίεση όσον αφορά την ε, επικουρικότητα και τις επιδοτήσεις θα είναι πάρα πολύ ε, ισχυρή. Διότι αυτό το οποίο δεν θέλουν να ξαναδούν οι κυβερνήσει είναι θεσμικά όργανα να αποτυγχάνουν, τον οποίο τη διαχείριση ως αποτυχία δεν μπορούν να αναλάβουν και να αποτελεσματικά να αντιμετωπίσουν. Να είμαι συντομότερος λέτε. Πολύ καλά. Εντάξει. Ευχαριστώ. Νομίζω ουσιαστικά κάλυψα τα περισσότερα ερωτήματα. Μη, ε, ε, και τελευταία τώρα. Ευρωπαϊκή Ένωση ε, απέναντι ή αντίθετη στην, στη ΣΥΠΑ. Είναι ένα θέμα εδώ. Πρέπει στην ΕΕ να κάνουμε αυτές τις ρυθμιστικές αλλαγές. Πρώτα και κύρια για το δικό μας συμφέρον. Θέλουμε οι δικές μας ευρωπαϊκές τράπεζες να, έχουν καλύτερα, να είναι καλύτερα εξοπλισμένες με κεφάλαια, ποιοτικά να μπορούν να δράσουν καλύτερα, να αντιμετωπίζουν καλύτερα τους κινδύνους, ε, να προστατεύονται καλύτερα. Αλλά αυτό δεν επαρκεί, σωστό, διότι δεν θέλουμε να βρεθούμε σε μειονεξία, σε μειονεκτική θέση όσον αφορά τον ανταγωνισμό με άλλους. Γι' αυτό εδώ, σε σχέση με τις ΗΠΑ, δόθηκε μεγάλη προώθηση, τεράστια προώθηση στις μεταρρυθμίσεις και τώρα βρίσκονται στην νομοθετική ρύθμιση. Δεν εγκατέλειψαν την ιδέα μεταρρύθμισης ε, του χρηματοοικονομικού ε, συστήματος τους, Όλες οι προτάσεις ε, προέρχονται από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο Οικονομικών. Θα δούμε τι θα γίνει λοιπόν ε, μέχρι του χρόνου. Θα, θα πρέπει να έχουμε μια διαδικασία που θα βαίνει εκ παραλίλου από πλευρά μα. Πρέπει να θυμόμαστε όμω ότι είναι προ το συμφέρον μα να μεταρρυθμίσουμε το σύστημα εμεί οι Ευρωπαίοι. Εντάξει, τελείωσα κυρία Πρόεδρε. Σίγουρα θα έχετε και άλλες ευκαιρίες να ο κύριος Τροσκάν. Συγγνώμη, αλλά θα... Με συγχωρείτε, θα μιλήσω αγγλικά. Σε σχέση με αυτό που είπε ο Μάριο για τη ΣΥΠΑ και την Ευρώπη και τα λοιπά. Ένα στοιχείο εδώ είναι μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση και καλύτερης ποιότητας κεφαλαιοποίηση. Όμως, αυτό που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι το ερώτημα του υπερβολικά μεγάλο για να αποτύχει. Δεν έχει να κάνει μόνο με το μέγεθος αλλά και με την έλλειψη διαφοροποίησης. Μπορεί να μιλάμε δηλαδή για ένα μικρότερο ίδρυμα, αλλά λόγω της έλλειψης διαφοροποίησης μπορεί να είναι πολύ πιο επικίνδυνη η πτώχευσή του. Ένα δεύτερο θέμα. Η δομή της βιομηχανίας στη ΣΥΠΑ, στην Ευρώπη και ενδεχομένως και στην Ιαπωνία ή αλλού διαφέρει. Δεν ισχύουν οι ίδιοι κανόνες, δεν υπάρχει ο ίδιος ανταγωνισμός. Γι' αυτό αν έχουμε μια παγκόσμια λύση όπως προτείνω εγώ αυτό δεν θα σημαίνει ότι θα ισχύουν ακριβώς οι ίδιοι κανόνες παντού, γιατί τότε κάποιος ε, θα ευνοείται περισσότερο από άλλους. Αυτό αφορά και τις αγορές συναλλάγματος. Για το δεύτερο σημείο, αν το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ θέλει να γίνει μια μεγάλη ρυθμιστική αρχή, μα είναι. Αυτή είναι η βασική δουλειά μας. Ο έλεγχος η παρακολούθηση. Το Δέλτα ΝΙΤΑΦ δημιουργήθηκε προκειμένου να συγκεντρώνει τις ρυθμιστικές αρχές, να προτείνει νέες ρυθμίσεις, τις οποίες θα εφαρμόζετε εσείς και εμείς στη συνέχεια επανερχόμαστε για να δούμε αν εφαρμόστηκαν σωστά οι κανόνες. Άρα λοιπόν, κατά βάση, Είμαστε ένας οργανισμός αφοσιωμένος στην, στον έλεγχο, την παρακολούθηση. Πέρα από τη βοήθεια και τα λοιπά που συμβαίνει σε έκτακτες περιπτώσεις. Όμως, ισχύει επίσης ότι μέχρι στιγμής το Δέλτα Νιτάφ κατανοούσε την, τον έλεγχο ως μάκρο έλεγχο, μακροοικονομικό έλεγχο. Το πρόβλημα είναι ότι χρειαζόμαστε έναν οργανισμό που θα λειτουργεί μακροοικονομικά, αλλά και κάτι που θα λειτουργεί σε επίπεδο χρηματοοικονομικό, χρηματοπιστωτικό. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει η εντολή του ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ να διευρυνθεί έτσι ώστε να καλύπτει και αυτή τη μακροοικονομική, το μακροοικονομικό έλεγχο για την κυρία Φερέιρα και τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου. Νομίζω ότι θα πρέπει να επεξεργαστούμε αυτή την ιδέα. Ας υποθέσουμε ότι σε πέντε ή δύο ή δέκα χρόνια έχουμε μία νέα κρίση, όχι όμοια, αλλά αρκετά παρόμοια. Είναι μια πιθανότητα αυτή. Θα ήταν υπερβολικά αισιόδοξο να πιστεύουμε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία τέτοιου είδους κρίση στο μέλλον. Εγώ πιστεύω ότι θα ήταν πολύ δύσκολο για τα εθνικά κοινοβούλια να επανέλθουν και να ξαναπροσφέρουν χρήματα για τη διάσωση των τραπεζών. Δεν θα το, επιστρέψει, δεν θα το επιτρέψει η κοινή γνώμη θα πούνε ότι το κάναμε μια φορά για να σώσουμε τις τράπεζες, αλλά δεν θα το ξανακάνουμε. Ειδικά αν δείτε και την κατάσταση στον τραπεζικό τομέα σήμερα. Άρα, εφόσον υπάρχει η πιθανότητα μελλοντική κρίσης και αν όντω πιστεύουμε ότι θα είναι πολύ δύσκολο να απευθυνθούμε για δεύτερη φορά στους φορολογούμενους, τότε θα πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας τους πόρους για να αντιμετωπίσουμε τότε το πρόβλημα. Και όπως είπε και ο Μάριο, θα χρειαστούν κάποιοι πόροι που θα πρέπει να προκύψουν και από συνεισφορά του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Οι G20 ζήτησαν από το Δέλτα Νιτάφ να εξετάσει τέτοιου είδους περιπτώσεις και εξετάζουμε όλες τις πιθανές λύσεις. Όμως το πρόβλημα είναι ότι όλοι δεν έχουμε τους ίδιους στόχους. Αν κάποιος ζητάει φόρο που να προωθήσει μια ηθική ανάπτυξη, καλός, αλλά αυτό δεν μπορεί να βοηθήσει σε περίοδο κρίσεων. Και δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα από κάποιο τέτοιο φόρο για την αντιμετώπιση κρίσεων. Θα μπορούσαμε βεβαίως να πούμε ότι ένα μερίδιο αυτών των χρημάτων θα αφορά την ηθική ανάπτυξη, άλλο για τη διάθεση των τραπεζών. Πάντως δεν θα μπορούσε να... Πάντως σε κάθε περίπτωση αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μόνο μία φορά, όχι δύο. Γι' αυτό το λόγο ούτε και αυτό είναι εύκολο και επομένως συνεχίζουμε να εξετάζουμε προτάσεις. Τώρα, το ερώτημα για το ευρώ πάντα είναι δύσκολο να κάνουμε προβλέψεις. Ο Κέινς είχε πει ότι οι προβλέψεις είναι δύσκολες, ειδικά να αφορούν το μέλλον. Υπάρχουν κάποια νομίσματα που είναι υποτιμημένα, ειδικά στην Ασία, ειδικά το κινέζικο RMB Νομίζω ότι η κατάσταση θα εξελιχθεί αργά αλλά θα εξελιχθεί. Βέβαια, εγώ λέω ότι ένα νόμισμα είναι υποτιμημένο. Αν ήταν περισσότερο υπερτιμημένο, τότε θα μειώνονταν κάποια προβλήματά μας. Όμως, δεν μπορούμε να πιστεύουμε ότι όλα τα προβλήματά μας θα μπορούσαν να λυθούν με αλλαγή των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Δεν μπορούμε δηλαδή να κρυφτούμε πίσω από αυτό το πρόβλημα και να διαφορήσουμε για προβλήματα όπως το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας, η παραγωγικότητα κτλ. Ναι, είναι σημαντικό θέμα οι ισοτιμίες, αλλά δεν είναι το μοναδικό ή το πιο σημαντικό. Και το τελευταίο ερώτημα του κυρίου Μπούλμαν. Με δύο τρόπους μπορώ να δω αυτό το ερώτημά σας. Λέτε, θα κάνουμε κάτι ή όχι. Σας λέω ξανά ότι για πρώτη φορά συνεργαστήκαμε τόσο πολύ. Τα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της κρίσης ήταν σε σύγκριση με πολλές δεκαετίες μοναδική περίπτωση που είχαμε εξελίξεις που βασίστηκαν στην πολιτική. Είχαμε το πακέτο κινήτρων, το ΔΝΤ ε, ζητούσε διαφορετικές παρεμβάσεις ίσως, αλλά εν πάση περιπτώσει για πρώτη φορά είχαμε τόσο μεγάλη κρατική παρέμβαση. Βεβαίως, το ερώτημα είναι τι θα κάνουμε από την άλλη πλευρά τώρα με την αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αυτό το ερώτημα παραμένει και με ενδιαφέρει και εμένα. Όμως, ας μην είμαστε υπερβολικά απεσιόδοξοι. Δεν είχε ξανασυμβεί τόσοι ηγέτες να λάβουν την ίδια απόφαση να χρησιμοποιήσουν τα δημόσια οικονομικά για να αποφύγουν τον κρεμό. Πρέπει λοιπόν να εξάγουμε τα διδάγματα των δύο τελευταίων ετών, που είναι οι αγορές λειτουργούν καλά, χρειάζονται μεγαλύτερη, καλύτερη ρύθμιση, όμως όποτε χρειαστεί μπορούν τα κράτη να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα. Νομίζω ότι αυτό είναι το τελικό συμπέρασμα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ακούσουμε λίγες παραπάνω ερωτήσεις αυτή τη φορά. Αν πρόκειται κάθε φορά οι απαντήσεις να κρατάνε δέκα λεπτά. Και δεν το λέω ως επίκριση αυτό για την αλήθεια ότι ακούσαμε πολλές ερωτήσεις. Ο κύριος Παλτασάρη από την Ιταλία θα πάρει τώρα το λόγο. Ε, Um, um, um, Παρακαλώ, μην είστε πολύ μακροσκελή στην παρέμβασή σας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τζάγκικ και τον κύριο Στάσκα, όχι μόνο για την πρωινή τους παρέμβαση, που έβριθε ενδιαφερόν των σημείων, αλλά που έμειναν λίγο περισσότερο μαζί μας μετά την ομιλία, αντίθετα με αυτά που έκαναν κάποιοι ομιλητές Έχω μόνο ε, δύο απλές ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά την διεθνή χρηματοστητική αρχιτεκτονική. Η δεύτερη αφορά το ρόλο της Ευρώπης. Αυτές οι προσπάθειες να σχεδιαστεί η νέα διεθνής αρχιτεκτονική είναι κάτι που χρειάζεται, είναι κάτι θετικό όμως δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο ποιες είναι οι οικοδομικές εταιρείε και ποιος είναι ο τελικός ιδιοκτήτης του κτηρίου που θέλετε να φτιάξετε. Το ερώτημα είναι αυτό. Αν η κρίση έχει τρεις βασικές ρίζες. Η μία από αυτές. Η πρώτη είναι η πραγματική ανισορροπία που υπάρχει στην παγκόσμια οικονομία, κυρίως μεταξύ ΙΠΑ και Κίνας πλεόνασμα αποταμιεύσεων, πλεόνασμα ε, κατανάλωσης. Δεύτερον, η έλλειψη κανόνων για τις χρηματοστικές αγορές. Άρα δημιουργούνται τέτοιες φούσκες οδοσκοπικές. Τρίτο θέμα είναι η έλλειψη governance, διακυβέρνησης. Άρα η προσπάθεια όσον αφορά τη διεθνή αυτή αρχιτεκτονική, χρηματοστατική, τη διεθνή χρηματοστατική αρχιτεκτονική, κινδυνεύει να μην μπορεί να αντιμετωπίσει την επόμενη διεθνή κρίση αν εν τω μεταξύ δεν υπάρχει πραγματική επανισορρόπηση και η νέα διακυβέρνηση, η governance. Δημιουργήσαμε ένα είδος Frankenstein. Μια αγορά Frankenstein που εκφράζει όχι τη χρεοκοπία της αγοράς αλλά τη χρεοκοπία του κράτους. Και γιατί είναι, έχει τη μορφή Φραγκενστάιν. Διότι αντιληφθήκαμε την παγκοσμιοποίηση σαν ελεύθερη ανταλλαγή εμπορευμάτων και υπηρεσιών μέσω του ΠΟΕ, όπου οι ποσότητες μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα, αλλά οι τιμές σε μεγάλο βαθμό αποφασίζονται από μια πολιτική απόφαση που λαμβάνεται στο Πεκίνο μέσω του pegging του κινέζικου γιουάν έναντι του δολαρίου, της οστιμίας αυτής. Αυτός ο Φράγκενστάιν λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο, θα τεθεί υπό έλεγχο, γιατί μπορεί να μας ξεφύγει από τον έλεγχο, από τα χέρια μας, όπως φαίνεται. Αυτή είναι η ρίζα της παγκόσμιας ανισορροπίας. Να έχουμε ακριβώς το να συμμετέχουν η Κίνα και άλλες χώρες της Ασίας την ελεύθερη συναλλαγή εμπορευμάτων και υπηρεσιών, αλλά αυτές να έχουν την δυνατότητα να αποφασίζουν ποιες είναι οι τιμές. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η χρηματοδοτική αρχιτεκτονική διεθνής θα πρέπει να ενταχθεί σε μια νέα governance που ξεκινά από ένα λέω Bretton, Bretton Woods. Διαφορετικά είναι δύσκολο να καταλάβουμε μετά την αρχιτεκτονική που χρησιμοποιείται με το πρόγραμμα AutoCAD και σχεδιάζεται αυτό το αρχιτεκτόνιμα, η οικοδομική εταιρεία που υπολογίζει τον Αγίο Σκυρόδεμα και το Χάλιβα, ποιο θα είναι και ποιο θα είναι ο τελικό ιδιοκτήτη του ακινήτου που θα είναι η νέα διακυβέρνηση, η νέα governance. Ποιο είναι ο ρόλο τη Ευρώπη. Ο ρόλο τη Ευρώπη είναι σημαντικό σίγουρα αλλά αυτή τη φορά είναι αδύναμη η Ευρώπη σε αυτή τη φάση. Διότι υπάρχει ένα πρόβλημα θεσμικής βάσης ευρωπαϊκής. Αυτό το δείχνει και η συνάντησή μα. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κυβέρνηση είναι υπόλογη σε εθνικέ κυβερνήσεις. Άρα δεν είναι πολύ ενδιαφέρον να υπάρχει συνομιλία με τα Εθνικά Κοινοβούλια ή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτός είναι ο κόμβος ο θεσμικός που πρέπει να μας οδηγήσει στο να δημιουργήσουμε όχι μόνο την Ευρωπαϊκή Αρχή Εποπτείας, αλλά κυρίως τα, τις Ηνωμένε Πολιτείε Ευρώπης, που φαίνεται μια ουτοπία, αλλά νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο είναι κάτι κατεπήγον. Η γερουσία της Ιταλίας και η δική μου επιτροπή των οικονομικών ολοκληρώνει μια έρευνα που διεξάγεται όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή. Ακριβώς αυτό το θέμα έχει κάτι που θα υποβληθεί στο Κοινοβούλιο και στην Ιταλική κυβέρνηση αυτή η έκθεση, αλλά ίσως να είναι κάτι που να ενδιαφέρει επίσης και τη συζήτησή μας σε αυτό το πλαίσιο. Η τελευταία ακρόαση θα είναι η τελική ακρόαση με την παρουσία του Επιτρόπου Μισελ Μπαρνιέ. Σε αυτή την έρευνα λοιπόν τι διαφαίνεται. Ένα σημείο σημαντικό που κατά την άποψη της Ιταλικής Γερουσίας θα πρέπει να ε, εξεταστεί εξονυχιστικά. Δηλαδή, έχουμε από τη μία πλευρά τον κίνδυνο να έχουμε ευρωπαϊκή αρχή, ευρωπαϊκές αρχές που είναι αυτοδύναμες αν θέλετε και αυτοελεγχόμενες και από την άλλη πλευρά με μια πολιτική που αντί τελευταίο σημείο αναφορά να είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, αυτές οι ανεξάρτητες αρχές να ε, δημιουργούν ένα μείγμα που παρεμβαίνει, ε, να δημιουργείται ένα μείγμα που παρεμβαίνει σε αποφάσει των εξαρτήτων αρχών. Αυτό το είδε ότι υπάρχει σαν κίνδυνο η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού, της, Ευρωπαϊκής, της Ιταλικής Γερουσίας, συγγνώμη. Και είναι κάτι το οποίο επιλύεται αλλά ακόμα δεν έχει λυθεί. Χρειάζεται να υπάρχουν ανεξάρτητες αρχές όπως έλεγε ο κύριος Ντράγκε που θα έχουν και το ρόλο της εποπτείας και το ρόλο να προειδοποιούν και το ρόλο να επιβάλλουν κυρώσεις. Και αυτές οι αρχές, οι ανεξάρτητες, θα πρέπει όμως να είναι υπόλογες στην, ε, στο Κοινοβούλιο το Ευρωπαϊκό και στην κυβέρνηση την Ευρωπαϊκή, διότι αυτό είναι ο κανόνας της δημοκρατίας. Και μια τελευταία ανησυχία, Πρόεδρε. Από αυτή την έποψη, λοιπόν, των πραγμάτων, προφανώς ο χρονισμός, το timing της αναδιάθρωσης της θεσμικής, της διεθνούς και της ευρωπαϊκής χρειάζεται χρόνο για πολιτικές ζημώσεις, ε, για συνένεση και ποια είναι η ανησυχία μου ότι οι χρόνοι που προβλέπονται για την ε, είναι πολύ σύντομοι από τους αναγκαίους για να δημιουργηθούν θεσμοί που θα είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν την κρίση και η ανάκαμψη που ευτυχώς ξεκινά αν βασίζεται στις ίδιες τρεις ρίζες που δημιούργησαν την προηγούμενη κρίση ε, ε, ε, ίσως βλέπουμε να ξαναφορτίζεται ένα νέο ελωτήριο κρίσης που θα σωρεύσει τις ίδιες εντάσεις και τάσεις σε λίγα χρόνια. Έχουμε πρόκληση μεταξύ χρόνου που χρειάζεται για πολιτική αναδιάρθρωση και θεσμική αναδιάρθρωση και τους χρόνους που απαιτείται για να βγούμε από την κρίση. Ο πρόεδρος ασχο... Βέβαια, η πρόεδρος ε, φροντίζει και για τους χρόνους της συνεδρίασής μας. Λοιπόν, Χρειάζεται αναδιάθρωση σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο των θεσμών. Χρειάζεται και χρόνο, περισσότερο χρόνο για αυτό από ό,τι για να βγούμε για την κρίση. Και αυτή η διαφορά των χρονισμών ίσως μας οδηγήσει σε νέες συνθήκες που οδηγήσουν σε νέα διεθνή κρίση. Χωρίς να έχουμε ακόμα δημιουργήσει τους ανεστέους φορείς και τα αναγκαία μέσα για την αντιμετώπιση των μελλοντικών κρίσεων. Αυτά ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ λέει Πρόεδρος. Δεν θα μπορέσω να σας δώσω τόσο χρόνο να μιλήσετε και έχω ένα κουμπί που σα διακόπτω και από εδώ και πέρα ίσως θα πρέπει να το χρησιμοποιήσω. Επόμενος. Πασκάλ Κανβέν. Σας έχασα. Α, εκεί είσαστε. Έχετε το λόγο. Θα προσπαθήσω. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Η ερώτηση προς τους κυρίους Τροσκάν και Τράγκη. Μιλήσατε για τον επιθυμητό πληθυρισμό. Χτες ε, είχαμε και έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που ανέφερε τα σχετικά επιχειρήματα. Θα ήθελα όμως να ακούσω περισσότερα και από εσάς και να μας πείτε ποια είναι η απάντησή σας κύριε Στροσκάν στα όσα επιχειρηματολογεί η καπατάφα. Και κύριε Ντράγκη, ζητάτε ολοκληρωμένο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Όμως ε, δεν μπορούμε να το έχουμε αυτό αν υπάρχουν μαύρα τείχη εντός του συστήματος. Μέχρι σήμερα οι συμφωνίες που υπογράφονται στο ICD και στις διάφορες ε, διεθνείς συμβάσεις δεν αλλάζουν κάτι επί τόπου. Οπότε, ποια συγκεκριμένη πρόταση έχετε να κάνετε για την αλλαγή της κατάστασης. Η Βαρόνη Κόεν από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είμαι πρόεδρος της Επιτροπής της Βουλής των ε, Λόρδων που γράφει εκθέσεις για τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε κάνει πολλές εκθέσεις φέτος και μία αφορούσε στις 31 Μαρτίου τα παράγωγα. Γιατί συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Ντράγκη όσον αφορά τη σημασία των παραγόγων, ειδικά όσον αφορά τον swap για την ανταστάθμιση του κινδύνου αθέτησης των CDS. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Μπορούμε να συνδυάσουμε μια πιθανή ευρωπαϊκή λύση με αυτό με το οποίο καταλήγουμε σε διεθνές επίπεδο, γιατί κάτι διαφορετικό θα έθετε σε κίνδυνο την ε, η οικονομική σταθερότητα και επίσης ως εκπρόσωπος μιας χώρας που ζει από τις οικονομικές υπηρεσίες αλλά και η οποία επίσης χώρα όταν εγκρίνει νομοθεσία την εφαρμόζει όπως είπε και ο Μάριο Μόντι. Οπότε θα έχουμε πραγματικές συνέπειες. Άρα, μία πολύ ευθεία και απλή ερώτηση. Πότε πρόκειται να έχουμε αυτές τις παγκόσμιες λύσεις για να τις υιοθετήσουμε όλοι. Για παράδειγμα για τα παράγωγα. Φοβάμαι ειδικά μετά από αυτό που είπε ο κύριος Μπαρνιέ ότι θέλουν να είναι στην πρωτοπορία ότι οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα παράγωγα δεν θα συνάδουν με τις παγκόσμιες λύσεις. Ρωτάω λοιπόν πότε θα έχουμε κάποια παγκόσμια λύση έτσι ώστε να μπορούμε να τη συγκρίνουμε με τις ευρωπαϊκές αναλλακτικές και να μπορούμε να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε. Κύριε Ποδηματά. Thank Ευχαριστώ. Θα μιλήσω ελληνικά γιατί θέλω να είμαι ακριβής. Θα συνεχίσω λίγο την παρέμβαση του συναδέλφου του Ούντο Μπούλμαν και με αφορμή και τα σχόλια του κυρίου ε, Στροσκάν. Κάνουμε μεγάλη συζήτηση στην Ευρώπη και παγκοσμίω, κάναμε και εδώ σήμερα, ε, για το αν και κατά πόσο τα σημάδια ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι βιώσιμα, σταθερά έχουμε την αίσθηση ότι δεν έχουμε αναλύσει αρκετά δεν έχουμε επεξεργαστεί αρκετά τα αίτια αυτής της παγκόσμιας κρίσης που ξεκίνησε από τον χρηματοπιστωτικό τομέα από την αμερική και εξελίχθηκε γρήγορα σε οικονομική και ε, κοινωνική. Ε, κύριε στροσκάν καλέσατε τον ε, συνάδελφο να μην είναι απεσιόδοξος και να μην υποβαθμίζει τον συντονισμό που υπήρξε σε παγκόσμιο επίπεδο ε, για την ε, αντιμετώπιση της κρίσης παραμένει βεβαίως το γεγονός ότι αυτός ο συντονισμός ο αποτελεσματικός ήταν κατασταλτικού χαρακτήρα ε, και διαρωτόμαστε εδώ στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο εάν οι συζητήσεις που γίνονται και στις δύο πλευρές του ατλαντικού για την νέα αρχιτεκτονική του χρηματοπιστωτικού συστήματος για καλύτερους κανόνες και καλύτερη εποπτεία έχουν πραγματικά συνυπολογίσει τα αίτια αυτής της κρίσης και προχωρούν σε εκείνες τις προτάσεις που πραγματικά θα αποτρέπουν την επανάληψη τέτοιου είδους κρίσεων ε, στο μέλλον είπατε ότι χρειάζεται ασφαλώς μια καλύτερη ρύθμιση στις αγορές το ερώτημα είναι χρειάζεται απλώς μια καλύτερη ρύθμιση ή μήπως χρειάζεται μια άλλη ισορροπία και αυτό είναι ένα δίδαγμα που πρέπει να αντλήσουμε από την κρίση ανάμεσα στις αγορές και στην πολιτική. Ε, πριν από δύο τρεις μέρες υπήρχε ένα άρθρο στις financial times όχι σε κάποια κομμουνιστική ή σοσιαλιστική εφημερίδα που είχε τον τίτλο γιατί οι αγορές πρέπει να υποδεικνύουν πολιτική ε, στους πολιτικούς. Ε, επειδή λοιπόν εδώ στο κοινοβούλιο έχουμε την αίσθηση ότι ε, αυτά που συζητιώνται για την αναμόρφωση της αρχιτεκτονικής του παγκόσμιου αρχιτεκτονικού συστήματος δεν είναι αρκετά φιλόδοξα ε, ώστε να αποτρέπονται τέτοιου είδους κρίσεις στο μέλλον θα ήθελα το, σχόλιο σας επ' αυτού. δεύτερο ερώτημα πολύ σύντομο αγορά παραγόγων αναφέρθηκε ο κύριος ντράγκη αναφερθήκατε κι εσείς και ο κύριος μπαρνιέ. το ερώτημα είναι επειδή υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες ε, η αγορά των παραγόγων και ειδικά τα credit default swaps. Έχετε την εντύπωση με βάση τα στοιχεία που έχετε στη διάθεσή σας ότι έπαιξαν ρόλο στην επιδείνωση της δημοσιονομικής κατάστασης της Ελλάδας και τι είδους ρυθμίσεις νομίζετε ότι πρέπει να υπάρξουν σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο σε ό,τι αφορά ε, αυτού του είδους τα παράγωγα σε σχέση βεβαίως ε, με τα εθνικά ε, την σύνδεσή τους δηλαδή με εθνικές ομολογίες. και τρίτο και ολοκληρώνω κυρία πρόεδρε ε, κύριε στροσκάν επειδή δεν έχουμε συχνά την τιμή και τη χαρά να σας έχουμε μεταξύ μας ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω γνωρίζετε ότι γίνεται μια συζήτηση πολύ μεγάλη αυτή την περίοδο για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού νομισματικού ταμείου θα ήθελα λοιπόν νομίζω ενδιαφέρει όλους τους συναδέλφου να ζητήσω την αντίδρασή σας σε σχέση με αυτή την προοπτική εάν νομίζετε ότι χρειάζεται ε, η δημιουργία ενός τέτοιου οργανισμού για την ε, αρρωγή τη συνδρομή ε, χωρών μελών της ευρωζώνης με μεγάλες δημοσιονομικές δυσκολίες εάν θεωρείτε ότι θα υπήρξε αλληλοεπικάλυψη ανάμεσα σε ένα τέτοιο θεσμό και το, το, νομισματικό ταμείο τρίτον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 ναι, αλλά πιο ανεκτικοί. Ναι, είστε μέλος του Κοινοβουλίου και γνωρίζετε ποιοι είναι οι χρονικοί περιορισμοί, ενώ τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων δεν είναι τόσο συνηθισμένοι. Με συγχωρείτε που είμαι τόσο αυστηρή, αλλά έχουμε πάρα πολλούς που έχουν ζητήσει το λόγο. Η κυρία Γκριν από τη Σουηδία έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς στην Σουηδία μέχρι τώρα την κρίση την αντιμετωπίσαμε σχετικά καλά θα έλεγα. Ακόμα και αν ε, έχουμε υψηλότερη, δυσανάλογα υψηλή ανεργία. Όμως ε, σε γενικούς όρους καλά τα καταφέραμε. Είχαμε καταρχήν ήδη θέση εντάξει τα της οικονομίας μας και είχαμε δημιουργήσει εποπτικές αρχές, είχαμε και πλεονάσματα όσον αφορά τα δημοσιονομικά μας. Είχαμε συναγάγει συμπεράσματα από την κρίση της δεκαετίας του 90, ακόμα και αν ήταν πολύ σκληρά αυτά και ομάτα συμπεράσματα τα υιοθετήσαμε. Υπάρχει όμως και ένας άλλος παράγοντας, ότι έγκαιρα γυναίκες εμπλέξαμε στην αγορά εργασίας όλες τις εργασίες, σε όλες τις εργασίες και δράσεις ισότιμα συμμετέχουν οι γυναίκες για την αντιμετώπιση της κρίσης. Και όσον αφορά την περαιτέρω πορεία, πώς μπορούμε να βρούμε μια διέξοδο από αυτή την κρίση και πώς θα εργαστούμε μέχρι το 2020, τρία πράγματα πρέπει να τονίσουμε. Πρώτον, η οικονομία πρέπει να είναι εξισορροπημένη, να επιτευχθεί μια ισορροπία των πραγμάτων. Χρειαζόμαστε μια ε, τάξη πραγμάτων στα οικονομικά και χρειαζόμαστε εποπτεία, σε αυτές τις αγορές για να υπάρξει αυτή η σταθερότητα και να αντιμετωπίσουμε περιπτώσεις κρίσεων. Δεύτερον, περισσότεροι πρέπει να μπορέσουν να εργάζονται. Πλήρης απασχόληση πρέπει να είναι ένα σημαντικό στόχος. Αυτό ισχύει και για άνδρες και γυναίκες. Πρέπει να είναι ασφαλείς θέσεις εργασίες αυτές. Πρέπει να είναι αναβαθμισμένες υψηλής ποιότητας θέσεις εργασίας. Πρέπει να αποφύγουμε να έχουμε μια σπυροειδή εξέλιξη προς τα κάτω όσον αφορά τους μισθούς και την απασχόληση. Πρέπει αναβαθμισμένα να προσπαθήσουμε να εργαστούμε και να πετύχουμε τους στόχους μας. Η αγορά εργασίας είναι σημαντική υπόθεση. Δεν πρέπει όμως να ασκείται αρνητική ε, διάκριση όσον αφορά τους εργαζόμενους. Πρέπει παντού για την ίδια εργασία να καταβάλλονται ίδιοι μισθοί, ίσοι μισθοί. Η άλλη διάσταση είναι η κοινωνική διάσταση. Αυτό είναι εξίσου σημαντικό όσον αφορά την οικονομία. Διότι μόνο μέσα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας μπορούν ε, να εργαστούν αποτελεσματικά οι άνθρωποι. Η μέρημνα, η περίθαλψη των παιδιών, κοινωνικά σημαντικά θέματα. Είναι, ασφαλ... είναι θέματα πολύ σημαντικά για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Αυτά ήθελα να πω σας σοσιαδημοκράτησα από την Σουηδία. Ευχαριστώ. And Philippe Lambert. Thank you, Chair. Yes, Philippe Lambert. Questions, one for each of our uh, speakers. First, uh, to Mr. Uh, Strauss κάποιες ερωτήσεις για όλους τους ομιλητές. Καταρχάς για τον κύριο Στροσκάνα. Όταν μιλάμε για μακροοικονομικές ανισορροπίες, συχνά εννοούμε το, έλεγχο, το έλλειμμα του ισοζυγίου ή το έλλειμμα το δημόσιο. Όταν μιλάμε για Ευρώπη και Ηνωμένε Πολιτείε, θεωρείτε ότι το χάσμα μεταξύ εισοδημάτων και την αύξηση των φτωχών που εργάζονται είναι μια συνέπεια της κρίσης ή ήταν ένας από τους λόγους της κρίσης. Θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας σχετικά. Και προς τον κύριο Ντράγκη, εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, είμαι μηχανικός και σκέφτομαι απλά. Όταν εμπορεύομαι με κάποιον, μπορώ να κάνω ασφάλεια για αθέτηση υποχρεώσεων. Αν μπορώ να το κάνω αυτό, τότε γιατί χρειάζομαι τα CDS. Δεν ξέρω αν είμαι αφελής, αλλά μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό. Κάποιες ακόμη ερωτήσεις θα ακούσουμε τώρα. Συσμές από την Ολλανδία, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ουσιαστικά θα ήθελα να συνεχίσω σε σχέση με την ερώτηση που διατυπώθηκε όσον αφορά το ευρωπαϊκό κίνημα, την προσπάθεια των Ευρωπαίων να δημιουργήσουν ένα ευρωπαϊκό νομισματικό ταμείο από πλευράς τους. Τώρα, διακόπτεται κάπως ε, το θέμα αυτό, διακόπηκε. Όμως θα ήθελα τον κύριο Στοσκάν να ακούσω κάτι παραπάνω για αυτό το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Η Ευρώπη στον πολιτικό προβληματισμό εξεταζόμενη ίσως θα μπορούσε να καταφέρει να πετύχει αυτό το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο με τη βοήθεια και υποστήριξη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δεν βλέπετε ότι υπάρχει εδώ ένα εξαιρετικό μέσο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που θα ήταν το πιο κατάλληλο να υλοποιήσει αυτό το ρόλο και θα έπρεπε να υλοποιήσει αυτό το ρόλο στην Ευρώπη ώστε χρηματοοικονομικά προβλήματα να μπορούν να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά και να επιληθούν όσον αφορά τους πιο αδύναμους. Στην εισαγωγή σας εσείς κυρίες Τροσκάν είπατε πόσο σημαντικό είναι το θέμα της πολιτικής ηγεσίας, στεναρής πολιτικής ηγεσίας για την επίλυση, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Δεν θέλω τώρα πολιτικά να έχω μία τοποθέτηση, αλλά να μου πείτε ως ειδικό. Ποιε είναι οι ικανότητες και οι δυνατότητες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ως προς αυτό. Πώς κρίνετε εσείς την Ευρωπαϊκή Επιτρα... στην Επιτροπή για ένα... τη δημιουργία ενό τέτοιου θεσμικού οργάνου και την διαχείρισή του. Ή βλέπετε και θεωρείτε κάποιου κινδύνους ε, να διαγράφονται. Όσον αφορά την πρόθεση τη δημιουργία ενό τέτοιου θεσμικού οργάνου του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου, με καλέ προθέσει βέβαια, αλλά όταν θα δημιουργηθεί να είναι μεγαλύτερη κίνδυνη από ότι οι καλέ προθέσει που το δημιούργησαν. Ευχαριστώ. Αυτό ήθελα να πω. Και να προσθέσω εδώ και την εξή παρατήρηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πολυσχηδής προβληματισμός για το μέλλον της ε, οικονομίας και το scaling και το πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν ε, τα προβλήματα των τραπεζών και να υποπτεύονται οι τράπεζες. Πολλές τράπεζες είναι too big to fail, υπερβολικά μεγάλες για να αποτύχουν, αλλά και too big to help, υπερβολικά μεγάλες για να βοηθηθούν λόγω τεραστίων κονδυλίων. Προς την κατεύθυνση αυτή σκέφτεται να κινηθεί η κυβέρνηση Ομπάμα. Τουλάχιστον θεωρεί ότι οι μικρότερες ε, ε, τράπεζες θα είναι εκείνες οι οποίες θα πρέπει να βοηθηθούν ε, και όχι οι μεγάλες. Αυτό τι σημαίνει. Οι τράπεζε θα πρέπει να βρίσκονται σε αναλογία με το μέγεθο τη χώρα και το μέγεθο ε, τη ίδια ε, τη τράπεζα. Για παράδειγμα, σε σχέση με την Ολλανδία ή Γερμανία, πώ θα μπορούσε αυτό να ισχύει. Συμμερίζονται αυτή την ε, άποψη οι αγορητέ ότι τέτοια προσέγγιση μπορεί να είναι βλαπτική για την λειτουργία μια αγορά, τη ευρωπαϊκή εδώ αγορά. Επειδή ιδιαίτερα μικρότερε χώρε θα είχαν μικρότερε τράπεζε και έτσι θα είχαν λιγότερα πλεονεκτήματα και λιγότερες δυνατότητες ανταγωνισμού στον, στην ανταγωνιστικότητά τους. Πώς θα μπορούσατε να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Ρόμπερτ Γκέμπελς είναι επόμενος που έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο Ντομινίκ Στρόσκαν καλά μας επέστησε την προσοχή στο γεγονός ότι οι ίδιοι κανόνες από την μία πλευρά του Ατλαντικού και την άλλη πλευρά του Ατλαντικού δεν έχουν τις ίδιες συνέπειες. Έχουμε το παράδειγμα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας που χρηματοδοτείται κατά δύο τρίτα μέσω τραπεζικών πιστώσεων, ενώ στις Ηνωμένε Πολιτείε είναι λιγότερο από ένα τρίτο. Όσον αφορά αυτό το θέμα, θα ήθελα να γνωρίζω αν οι ελπίδες που ο Μάριο Ντράγκη και ο κ. Σκάν ε, δίνουν στις εργασίες της Επιτροπής της Βασιλείας όσον αφορά αυτό το θέμα ε, είναι βάσιμες. Εγώ από ό,τι γνωρίζω για τη Βασιλεία 2, η Βασιλεία 2 δεν έχει εκτελεστεί ακόμα από τους Αμερικανούς, ενώ εδώ μιλάμε για τη Βασιλεία 3 και μιλάμε μόνο για υποχρεώσεις για τις Ευρωπαϊκές Τράπεζες με δεχόμενη στρέβλωση του ανταγωνισμού που συνεπάγεται αυτά που σχολίασε ο Ντομινίκ Στροσκάν. Και άλλη παρατήρηση προς τον Μισελ Μπαρνιέ που δυστυχώς απουσιάζει που μας την έκκληση και παραθέτω ανάπτυξη πιο πράσινη, πιο δίκαιη, πιο ισότιμη. Τέλος παράθεσης. Ε, γνωρίζω ότι είναι της μόδας να μιλάει κανείς για μια ανάπτυξη πιο πράσινη. Ενώ οι καλύτερε εκτιμήσει μα λένε ότι θα έχουμε 2 εκατομμύρια θέσει πράσινε μέχρι το 2020, ενώ έχουμε 23 εκατομμύρια ανέργου στην Ευρώπη. Θα πρέπει να επενδύσουμε και στι παραδοσιακέ βιομηχανίε για να δημιουργήσουμε θέσει απασχόληση και να δούμε πραγματική ανάπτυξη. Εγώ προσωπικά θα ικανοποιούμουν με μεγαλύτερη ανάπτυξη, είτε πράσινη είτε όχι και πιο δίκαιη, πιο ισότιμη ανάπτυξη μπορώ να κάνω τίποτα. Το πρόβλημα δεν είναι η πιο δίκαιη ανάπτυξη, η πιο ισότιμη ανάπτυξη. Το πρόβλημα είναι η κατανομή των καρπών της ανάπτυξη που πρέπει αυτή η κατανομή να γίνει πιο δίκαιη και πιο ισότιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα επανέλθω στους ομιλητές μας για να δώσουν κάποιες απαντήσεις. Να σας γνωστοποιήσω ότι έχουμε άλλους οκτώ ομιλητές που περιμένουν να πάρουν το λόγο. Σας παρακαλώ προσπαθήστε να είστε όσο πιο λακωνικοί γίνεται για να έχουμε το χρόνο για έναν τελευταίο γύρο. Κύριε Κράγκη, για μία ακόμη φορά έχετε το λόγο πρώτος. Κυρία Πρόεδρε, δεν μπορεί να πετύχει κανείς και τα δύο. Να έχει κανείς πολύ, πολλές ερωτήσεις που βάλλονται και πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να απαντηθούν. Σας ζητώ συγγνώμη. Επίοικια. Στο πρώτο τμήμα της πρώτης ερωτήσεως να απαντήσω. Ποια είναι η μορφή της χρηματοπιστωτικής αρχιτεκτονικής που θα απορρεύσει από όλα αυτά. Είπα στην αρχή κάποια πράγματα. Ο επιμερισμός των εργασιών, η κατανομή των εργασιών που κάναμε με τον Ντομινίκ, τι μας λέει ότι η FSB σχεδιάζει τους κανόνες και το Εθνές Νομισματικό Ταμείο ασκεί την εποπτεία και οι εθνικές αρχές και οι νομοθέτες θα εφαρμόσουν τους κανόνες. Αυτό είναι ένα κομμάτι της αρχιτεκτονικής, του αρχιτεκτονήματος. Το δεύτερο τμήμα του αρχιτεκτονήματος αφορά τις, του φορεί που καθορίζουν διεθνεί προδιαγραφέ. Δηλαδή την Επιτροπή τη Βασιλεία στο αφορά σύστημα, το αντίστοιχο τη Επιτροπή Βασιλεία στο σύστημα ασφάλιση και έχετε και τι εποπτικέ αρχέ τη αγορά τα διάφορα SEC στη ΣΥΠΑ, FSA στο Ηνωμένο Βασίλειο κλπ. Commission Bancaire στη Γαλλία και όλοι αυτοί ομαδοποιούνται σε διεθνή φορεία, φορέα των IOSCO. Και έχετε και τους λογιστές, την EISB. Τι είπαν οι G20. Καλώς όλοι αυτοί οι φορείς θα πρέπει κάπως να συντονιστούν από την FSB. Και αυτό απεδείχθη μια χρήσιμη απόφαση. Εδώ ίσως να μεροληπτώ, διότι επιταχύνθηκε το πρόγραμμά μας τρίτο τρόπος τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Αυτή είναι η αρχιτεκτονική που έχουμε τώρα και πιθανότατα αυτή θα είναι η τελική αρχιτεκτονική. Εδώ θα σταματούσα όσον αφορά το χρηματοπιστωτικό τμήμα, τις χρηματοπιστωτικές αγορές και όσον αφορά το τραπεζικό τομέα. Ο Ντομινίκ θα αναφερθεί στην αρχιτεκτονική δομή των διεθνών εποπτικών φορέων. Στο δεύτερο ερώτημα έρχομαι. Τι κάνουμε για τις νομοθεσίες που δεν είναι συνεργάσιμες. Πολύ δουλειά έγινε ξεκινώντας με τη χάρτα της FSB. Τα μέλη της FSB δεσμεύτηκαν να ηγηθούν δίνοντας το παράδειγμα. Δηλαδή να συμμορφώνονται με τις διεθνές, διεθνείς προδιαγραφές και να κάνουν τι καλύτερο μπορούν ούτως ώστε τα να, να ασχολούνται με μη ε, συμμορφούμενες νομοθεσίε όσον αφορά τι διεθνεί προδιαγραφέ. Ξεκινήσαμε αυτό το μήνα μια πρωτοβουλία να συμφωνήσουν όλε οι νομοθεσίε με τι διεθνεί χρηματοστητικέ προδιαγραφέ και να εντοπίσουμε και να δακτυλοδεικτήσουμε τι νομοθεσίε εκείνε που δεν συμμορφώνονται και να του βοηθήσουμε να συμμορφωθούν. Πού εστιάζεται η προσπάθεια, σε συμμόρφωση με διεθνείς προδιαγραφές για τη συνεργασία και τη συμμόρφωση ε, στους τομείς εποπτείας και ελέγχου τους διεθνείς. Η FSB για ε, τις νομοθεσίες εκείνες που δεν συμμορφώνονται και δεν συνεργάζονται στον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών θα καλέσει τις νομοθεσίες να ξεκινήσουν διάλογο για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε κατά πόσο συμμορφώνονται και να εντοπίσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορεί αυτή η συνεργασία τους να βελτιωθεί. Είναι ένας τομέας στον οποίο πρέπει να κινηθούμε μαζί με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα. Και αυτοί οι δύο εντός των πλαισίων που μπορούν να κινηθούν, εντός της χάρτας τους. Για τα OTCs ε, σας ευχαριστώ πολύ για την τοποθέτησή σας και την δήλωσή σας. Όπως είπατε συμφωνούμε απόλυτα και αυτό που μπορώ να πω απαντώντας στο ερώτημά σας πότε μέχρι τον Οκτώβριο το FSB θα έχει μια πρόταση σχετικά με τις προδιαγραφές ε, που τα CCPs ή οι διάφοροι φορείς που συμμετέχουν θα χρησιμοποιήσουν για να προχωρήσουν και ποια προϊόντα, παράγωγα προϊόντα θα πρέπει να τυποποιηθούν για να υποστούν σε υποχρεωτικές απαιτήσει για κεντρικό έλεγχο, κεντρικό clearing. Όσο αφορά του οργανισμού συμψηφισμού, συμψηφισμού. Κοιτάξτε, Όσον αφορά τις ε, συζητήσεις στην Ευρώπη, πρέπει να δούμε ποιοι τελικοί εμπορικοί χρήστες θα πρέπει να εξαιρούνται από αυτές τις απαιτήσει, Θα πρέπει να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία. Και μπορώ να προβώ σε ένα γενικό σχόλιο πάνω σε αυτά. Όσο κινούμεθα προς εκτέλεση, υλοποίηση των όσων θα αποφασίσουμε στο τραπεζικό, στα OTC, στο too big to fail, όλα αυτά είναι πάρα πολλά Όσο προχωρούμε όμως, θα υπάρξουν θέματα επί των οποίων μπορούμε να συμφωνήσουμε ή εκεί που δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Και κάνουμε μια έκκληση σαν FSB. Παρακαλούμε, ας συγχωρούμε κάποια πράγματα. Τελικά προσπαθούμε να φτάσουμε σε τελική συνένεση όσον αφορά διάφορα ζητήματα και αυτός είναι ένας από αυτούς τους τομείς. Παράδειγμα, δεν θα ήθελα αυτό να είναι ένα σημείο στο οποίο να κολλήσουμε για μια γενική τυποποίηση των παραγόγων OTC. Δηλαδή το θέμα του ποιο τελικός εμπορικός χρήστης θα πρέπει να εξαιρείται από τις απαιτήσει. Τέταρτο θέμα για τα CDS, για τη συμβάση της τάθησης κινδύνου. Να ζητήσω συγγνώμη, διότι έπρεπε να, να λείπω για λίγο, ίσως να είναι τελής η απάντησή μου αυτό το λόγο, διότι απουσίαζα. Το ερώτημα είναι, ε, ήταν η ρίζα της ελληνικής κρίσης τα CDS, αυτό ήταν το ερώτημά σας. Το ερώτημα ήταν κατά πόσο επιδίνωσε το CDS ε, το πρόβλημα της ελληνικής κρίσης. Απάντηση. Όσον αφορά αυτό το θέμα, όπως και για το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, για αυτό το θέμα χρειάζομαι περισσότερο χρόνο, διότι είναι σημαντικό θέμα για διάφορους λόγους Και άλλο έθεσε το ίδιο ερώτημα, λέει η Πρόεδρος, στον ομιλητή. Καλώ. Θα απαντήσω και στις δύο ερωτήσει. Ας ξεκινήσω λοιπόν με την βάση. Ποια είναι η προϋπόθεση, η βασική υπόθεση. Ας εστιαστούμε επί της κρίσης εντός του πλαισίου του τι πετύχαμε μαζί τα τελευταία 15-20 χρόνια. Δημιουργήσαμε τη συνθήκη του Μάστριχτ. Δημιουργήσαμε το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Ο Ντομινίκ Στρόνσκαν ήταν Υπουργό Οικονομικών στη Γαλλία όταν έγινε αυτό. Με τη δημιουργία του ευρώ δώσαμε σταθερότητα στον τομέα της Ευρωζώνης. Είχαμε χαμηλό πληθωρισμό και χαμηλό κόστος χρηματοδότησης και πιο σημαντικό προστατευόμασταν από τις παγκόσμιες αναταραχές, από μια κρίση που αλλιώς δεν θα ξέραμε τι θα συνέβαινε στις διάφορες χώρες. Ξέρουμε ότι ό,τι λέμε και σκεφτόμαστε και αποφασίζουμε για την Ελλάδα αλλά και για άλλα πράγματα θα πρέπει να βασίζονται στο θέμα της σταθερότητας των τιμών και στη γενική χρηματοπιστωτική οικονομική σταθερότητα. Κάτι που πετύχαμε με πολύ ψηλό τίμημα. Τούτων λεχθέντων, τι είναι η ελληνική κρίση, είναι μια οικονομική κρίση. Πώς αντιμετωπίζουμε αυτή την κρίση. Εδώ έχουμε το, δάσκαλο για την αντιμετώπιση αυτών των κρίσεων. Αλλά οι πυλώνες της αντιμετώπισης της κρίσης αυτής της οικονομικής είναι εκ των προτέρων δεσμεύσεις, ανάληψη υποχρεώσεων και ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα με ανάληψη εκ των προτέρων υποχρεώσεων. Γιατί πρέπει να είναι εκ των προτέρων, διότι εκεί είναι τα μεγαλύτερα ωφέλη. Οι αγορές θα μειώσουν το spread, τα spreads αμέσως, αν έχουν αναλυφθεί εκ των προτέρων υποχρεώσεις, αμέσως. Θα πρέπει να είναι δομικής φύσεως. Από τη στιγμή που είναι ε, μέτρα που λαμβάνονται μια φορά η αγορά δεν τα λαμβάνει υπόψη. Λένε δεν είναι καλά τα μέτρα. Τρίτον, θα πρέπει να υπάρχει πολύ αυστηρό έλεγχο. Και τέταρτον, θα πρέπει να υπάρξει ταχεία εφαρμογή, πολύ ταχεία εφαρμογή. Και νομίζω ότι σε αυτή τη φάση αυτό είναι το σχέδιο. Αυτό έδειξε στην Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η συνεργασία με το Διεθνέ Ταμείο όλοι μαζί πίστηκαν ότι υπάρχουν αυτέ οι προποθέσει. Τώρα είναι θέμα εφαρμογή, εκτέλεση είναι εξίσου σημαντική, ακόμα πιο σημαντική από τον σχεδιασμό η εφαρμογή. Αν το κάνουμε αυτό, τα κάνουμε αυτά, έχω την πεποίθηση ότι οι αγορές θα είναι εκεί. Θα δανοδιοτήσουν, θα δώσουν τα αναγκαία ποσά, θα τα δανείσουν. Ας επιστρέψω σε ένα λεπτό στη δική μου προσωπική εμπειρία. Το 1991 η Ιταλία αντιμετώπιζε μια παρόμοια οικονομική κρίση και πολύ χειρότερη. Είχαμε ένα έλλειμμα όσον αφορά το ΑΕΠ πάνω από 11% Είχαμε ένα χρέος που αυξανόταν προς 100 και πάνω από 100%. Είχαμε υποβαθμιστεί επανειλημμένα, είχαμε πληθωρισμό περίπου 10% και η κοινωνική συνοχή είχε καταστραφεί από τα τελευταία υπολείμματα της τρομοκρατίας. Οπότε η κατάσταση ήταν πολύ χειρότερη. Βγήκαμε με προσαρμογές, οικονομικές αναγκές, έπρεπε να χρηματοδοτήσουμε, να χρηματοδοτήσουμε το βραχυπρόθεσμο χρέος για εκατοντάδες δισεκατομμύρια, δεκάδες δις ευρώ κάθε μήνα, για ένα χρόνο πρέπει να τα πληρώνουμε αυτά. Και δεν είχαμε εξωτερική δημόσια υποστήριξη σημαντική. Αν με ρωτάτε, α, ο καθένας μπορεί να το πετύχει αυτό χωρίς να δημιουργήσει ειδικού θεσμούς. Όμως, Πιστεύω ότι υπάρχει μια βασική διαφορά με αυτή την εμπειρία. Οι αγορέ τώρα είναι πολύ πιο τρομαγμένε μετά την, μετά την κρίση των Lehman Brothers από ό,τι κατά το παρελθόν. Είμαστε πιο ευαίσθητοι όσον αφορά το συστημικό κίνδυνο και οι κυβερνήσει δεν θέλουν να βλέπουν το χάο μπροστά του. Οπότε, ίσω να έχουμε προσωρινή ρευστότητα, ρε, ρευ... ανάγκε προσωρινές, έκτακτες ε, έτσι πρέπει να το δούμε σαν μια διευκόλυνση προσωρινή ρευστότητα. το IMF e όπως λένε οι Αμερικανοί σαν το κερασάκι στην τούρτα αλλά πρέπει να είναι έτοιμη η τούρτα εκ των προτέρων δηλαδή αξιόπιστες οικονομικές προσαρμογές θα πρέπει να έχουν εφαρμοστεί αυτό πρόθεσμα και θα σταματήσω επ' αυτού αλλά δεν αρκεί αυτό, δεν αρκεί διότι Έχουμε ακόμα χώρες με υψηλό χρέος και μικρή ανάπτυξη. Και αυτό δεν είναι καλό, διότι στο τέλος θα πρέπει να βρουν τα οικονομικά μέσα για να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Άρα πρέπει να αναπτυχθούν περισσότερο. Θα σταματήσω εδώ ε, και αν δεχτώ άλλες ερωτήσεις θα απαντήσω για το σχετικά το τι πρέπει να γίνει με αυτό. Τόσο αφορά το επόμενο ερώτημα για τα CDS. Έχετε δίκιο. Αρχικά δεν υπήρχαν CDS μέχρι τα τέλη, μέσα της δεκαετίας των 90. Και υπήρχε ασφάλιση των ε, πιστώσεων. Γιατί αυξήθηκαν τα CDS και δεν ασφαλίζουν ασφαλιστικές εταιρείες τις ίδιες πιστώσεις. Για πολλούς λόγους. Ένας από τους λόγους είναι ότι αν μια τράπεζα θέλει να ασφαλιστεί ε, ε, έναντι ενός συνόλου πιστώσεων περνάνε μέσω της διάβλου του CDS και όχι μέσω ασφαλιστικών εταιριών για λόγους που σχετίζονται με την δομή που έχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Ένας λόγος. Άλλος λόγος είναι ότι αυξήθηκαν τα CDS με, με έναν εντελώ ανεξέλεγκτον τρόπο, σε διαφορά, σε αντίθεση με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Το είδαμε αυτό. Οι ασφαλιστικές εταιρείε έχουν ένα ποσοστό φερεγγιότητας και πρέπει να έχουν κεφάλαιο έναντι των υποχρεώσεων και έναντι των ασφαλιστηρίων του είδαμε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείε τριπλού α όπως η AAG ε, μπορούσαν να δώσουν 400 δις ε, CDS χωρίς εγγύησεις. Οπότε αναπτύχθηκε ανεξέλεγκτα η αγορά. Τι να κάνουμε εδώ. Και εν μέρη το απάντησε αυτό. Είναι πολύ περίπλοκο το ερώτημα, βλέπετε θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ξανασχεδιαστούν οι συμβάσεις CDS ούτως ώστε να εξαιρεθούν οι ασφαλίσεις θα μπορούσε να γίνει πολύ δύσκολο. Το πρώτο βήμα είναι να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Δηλαδή, σε κεντρικό επίπεδο να ελέγξουμε το εμπόριο CDS. Αν το κάνουμε αυτό, θα έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια, πολύ μεγαλύτερη ορατότητα του τι κρύβεται πίσω από αυτά. Θα ξέρουμε ακριβώς ποιο είναι το καθαρό τμήμα και ποιο όχι. Πολλέ από τις εκτιμήσει και του υπολογισμούς ε, δεν είναι ακριβείς και θα ξέρουμε κάτι πολύ σημαντικό. Η εγγύηση, πώς γίνεται ο χειρισμός του, ε, των εγγυήσεων και πού βρίσκονται αυτές. Ο Ντομινίκ. Έχω άλλες δύο ερωτήσεις να απαντήσω. Η Πρόεδρος. Ε, ίσως ο κ. Στασκάν μπορεί να απαντήσει στις ερωτήσεις που παραλείψατε να απαντήσετε εσείς. Uh, κάποια σημεία. Πρώτα για την ιδέα νέας συμφωνίας, νέας ε, Bretton Woods. Μια θετική ιδέα να δημιουργηθεί κάτι καινούριο. Προφανώς ε, η Bretton Woods έχει 65 χρόνια παρελθόν και θα ήταν κάτι εκπληκτικό αν τίποτα δεν χρειαζόταν να αλλάξει. Όμως το ερώτημα είναι το πολιτικό κλίμα, ο πολιτικός περίγυρος μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κατέστησε εφικτή την διεξαγωγή αυτής της συνεδρίασης. Ε, δύο μήνες πήρε για τους εκπροσώπους, τους αντιπροσώπους των Bretton Woods για να συναυθεί αυτή η συμφωνία, αυτή η συνθήκη. Δεν είμαι σίγουρος αν σήμερα θα μπορούσε με τον ίδιο τρόπο να συντεθεί να διοργανωθεί κάτι παρόμοιο. Έχουμε και μεγαλύτερο αριθμό χωρών και εκπροσώπων, πράγμα το οποίο δυσχεραίνει τα πράγματα σε σχέση με αυτά που έγιναν πριν από 65 χρόνια. Γιατί όχι λοιπόν, όμως δεν είμαι βέβαιος, βλέποντας ας πούμε την σύνοδο της Κοπενχάγης και την προσπάθεια κατάληξη σε συμφωνία μεταξύ τόσου μεγάλου αριθμού εκπροσώπων τόσων πολλών χωρών, ο, ιωθός που επιλέξαμε μέσα στο ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι η επανεξέταση της εντολής. Να ξαναδούμε την εντολή και να ξαναδούμε πώς μπορούμε να είμαστε πιο επικοδομητικοί και αποτελεσματικοί, επεκτείνοντας τις δυνατότητες της δραστηριοποίησης μας, δράσης μας, αλλά όχι ξανασυντάσσοντας μια νέα συνθήκη. Γιατί πραγματικά φοβούμαι ότι κάτι τέτοιο θα απαιτούσε μεγαλύτερο χρόνο, μεγάλο χρονικό διάστημα. Όμως από την άλλη πλευρά, αν αλλάξω τώρα την παρέμβασή μου από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και μιλήσω σε ένας Ευρωπαίος πολίτης, δεν είμαι σίγουρος ότι αποβαίνει απόλυτα προς το συμφέρον του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να ζητήσει τη σύνταξη μιας νέας συνθήκης. Γιατί τότε το θέμα της εκπροσώπησης και της στάθμισης των ευρωπαϊκών χωρών θα ξανατεθεί. Και δεν είναι ένα θέμα στο οποίο θα ήθελα να επεκταθώ πολύ περισσότερο, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι αυτό θα μπορούσε να αποβεί προς το σαφές συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα πω τίποτα περισσότερο από αυτού. Δεύτερο, τώρα θα μιλήσω γαλλικά. Παραγατέ, ε, Ερώτηση επί του εγγράφου του κυρίου Μπλανσάρ, επικεφαλής οικονομολόγου του Ταμείου, το προηγούμενη εβδομάδα, για τους ε, λόγους της κρίσης. Πρόκειται για μια ερευνητική δημοσίευση που έδειξε που προσπάθησε να αναλύσει τι μάθαμε από την κρίση, από πού προήλθε η κρίση κτλ. Προκύπτουν διάφορα θέματα. Ένα από αυτά είναι και ο πληθωρισμός. Σίγουρα αυτό, αυτή η έρευνα έπρεπε να επικεντρωθεί και σε άλλα θέματα πέρα από το πληθωρισμό αλλά επειδή με ρωτήσατε για τον πληθωρισμό να πω ότι εγώ λέω παντού ότι μιλάμε για ένα νέο νομισματικό ταμείο, αν και παραμένει νομισματικό ταμείο. Και το δόγμα μας είναι ότι πρέπει συνεχώς να αγωνιζόμαστε κατά των πληθωριστικών πιέσεων γιατί ποτέ δεν έχουν θετικές επιπτώσεις. Βεβαίως τώρα τίθεται το ερώτημα του τι εκπροσώπηση χρειαζόμαστε, τι επίπεδο εκπροσώπησης Πρόκειται για ένα θεωρητικό ερώτημα και ανοιχτό ερώτημα. Και αυτό είναι ο ρόλος των κεντρικών τραπεζιών. Να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό. Γι' αυτό έχουν αυτή την θέση. Βεβαίως, στα ακαδημαϊκά, ακαδημαϊκά μάλλον στην ακαδημαϊκή συζήτηση, το συζητάμε όλο αυτό το θέμα, αλλά παρόλα αυτά το δόγμα του Δελτανιτά παραμένει αντιμετώπιση του πληθωρισμού. Και επανέρχομαι στα αγγλικά. Για το θέμα μιας καλύτερης εξισορρόπησης των πραγμάτων καλύτερης ισορροπίας από την οικονομία της αγοράς και των παρεμβάσεων. Είναι μια συνεχιζόμενη συζήτηση εμβρευστό. Παρ' όλα αυτά, το θέμα δεν είναι τόσο να πει κανείς και να εξετάσει και να πει τι είναι αυτά που γίνονται σήμερα για καλύτερη ρύθμιση των, του οικονομικου κόσμου, αν αυτά είναι φιλόδοξα ή όχι. Το θέμα είναι ποια είναι η ισορροπία των δυνάμεων, τι μπορεί να κάνει κανείς. Και όσο περισσότερο ασχολείται κανείς με την πολιτική, τόσο περισσότερο πρέπει να ασχοληθεί με θέματα ισορροπία, εξισορρόπησης ε, της εξουσίας. Έτσι λοιπόν, το μέτρο της φιλοδοξίας είναι δεδομένο και μεγάλο όσον αφορά την προσπάθεια εξισορρόπησης ε, των εξουσιών για τον σχεδιασμό ενός συστήματος καλύτερο από αυτό, από αυτό που έχουμε. Το θέμα είναι πού βρισκόμαστε σήμερα και τι θέλουμε να κάνουμε με το καινούριο νέο σύστημα. Υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά την ισορροπία των πραγμάτων και των εξουσιών στον πραγματικό κόσμο, στην πραγματική οικονομία. Δεν μπορεί κανεί να πει ότι δημιουργούμε, θα δημιουργηθεί ένα σύστημα μέσα στο οποίο, μετά από το οποίο δεν θα μπορεί να υπάρξει καμιά κρίση. Κάτι τέτοιο δεν θα ήταν, δεν είναι λογικό. Μετά, εργαζόμενοι πρέπει να επισκοπούμε και να κάνουμε μια αναδρομή σε σχέση με το παρεθόν, διότι τα πράγματα στο μέλλον θα είναι πλέον διαφορετικά. Ε, από την φύση των πραγμάτων δεν μπορεί κανείς να πει ότι θα αποφύγουμε οποιαδήποτε κρίση στο μέλλον. Το ελάχιστο που πρέπει να κάνουμε είναι να πούμε ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κάποια προβλήματα ώστε τέτοιου είδους κρίσεις να μην επαναληφθούν στο μέλλον, να μην μπορέσουν να επαναληφθούν. Αυτό είναι εκείνο το οποίο κάνουμε. Και σε σχέση με την πολιτική συνένεση που υπάρχει είναι δεδομένη ακόμα. Παρότι και, ε, ε, είπα στην ενακτήρια παρέμβασή μου ότι ήταν ισχυρότερη όταν βρισκόμαστε στην ακμή της κρίσης, στην πιο οξυμένη φάση της. Ο Μάριο και εγώ είμαστε παρόντες στη συνάντηση της λέσης των 20, G20. Δεν είναι κανένα μυστικό να πει κανείς ότι ήταν φοβισμένοι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Είναι πιο εύκολο να, αντιμετωπιστεί, να αντιμετωπίσει κανείς ε, φοβισμένους ε, ανθρώπους ε, ε, οι πολίτες. Και έτσι λοιπόν καλό ήταν ότι υπήρχε αυτός ο φόβος. Ε, τώρα, ποια θα είναι η έκβαση όσον αφορά την έκβαση της ισορροπίας των πραγμάτων μετά από δύο χρόνια δεν μπορώ να το προδικάσω. Ίσως ε, μπορεί να μην εμπλέκομαι πλέον σε τέτοια θέματα μελλοντικά. Όμως, παρότι δεν το πιστεύω, υπάρχει όμως πρόθεση των πραγμάτων και υπάρχουν κίνητρα και υπάρχει φιλοδοξία να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε αυτά τα πράγματα και μάλιστα η φιλοδοξία αυτή είναι υψηλού επίπεδου. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο σε αυτά τα οποία προανέφερε ο Μάριο. Μόνο μία παρατήρηση ίσως εδώ. Η πολύ μεγάλη αγορά είναι η αγορά των corporate CDS, credit default swaps. Κάποιε άλλε αγορέ δεν είναι τόσο μεγάλε. Είναι δύσκολο να ξέρει ακριβώς τι ακριβώ συνέβη. Θα πάρει χρόνο να, αναλυθεί το, να αναλυθούν τα συμβάντα των ε, τελευταίων εβδομάδων. Οι κινήσει για τα CDS δεν είναι τόσο σημαντικά όσο όταν κάναμε λόγο για τα CDS ε, λαμβάνοντας υπόψη τα corporate CDS. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Και τώρα για το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, όπως αποκαλείται. Θα ήμουν πολύ ικανοποιημένος ε, να μπορούσα να γνωρίζω περί τίνος πρόκειται ακριβώς και να το κατανοούσα ακριβώς. Άκουσα διαφορετικές ε, διατυπώσεις από διαφορούς ανθρώπους. Όλες έχουν κάποιο νόημα, αλλά εξαρτάται ποιαν εξετάζει κανείς. Αν κάποιος κάνει λόγο για την ιδέα ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να υπάρχει ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο Περιφερειακό που θα μπορούσε σε σχέση με χώρες όπως την Ουγγαρία, Λετωνία, Ρουμανία να βοηθήσει με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όμως η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να περνά μέσω αυτού του Αττικού Ταμείου και όχι μέσω των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού ε, Προϋπορισμού της ΕΕ. Αυτό εντάξει, αλλά αυτό δεν σχετίζεται τώρα σε σχέση με την Ελλάδα. Τώρα, μέσα στη ζώνη ευρώ, το θέμα αυτό το οποίο ανέφερε ο Μάριο, είναι πρώτα απ' όλα πάνω-πάνω. Το κύριο θέμα για την Ελλάδα δεν είναι αυτό. Τα θέματα είναι δημοσιονομικής πολιτικής ε, και αυτά πρέπει οικονομικά να αντιμετωπιστούν. Και σε σχέση με την ε, οικονομική πολιτική αυτά που πρέπει να γίνουν Πρέπει να είναι δημιουργική η δράση μας ε, από πλευράς ε, παρέμβασης θεσμικών οργάνων. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένα θεσμικό όργανο δεν θα μπορούσε να είναι χρήσιμο. Πρέπει να δούμε σε σχέση με την ε, ζώνη ευρώ να υπάρχει η δυνατότητα να διατεθούν κονδύλια, να βοηθηθεί μια χώρα. Θα υπάρχουν θέματα της ερμηνείας της συνθήκης. Δεν είναι πράγματα τα οποία μπορούν μια νυχτή να γίνουν για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ευρωζώνη με την Ελλάδα. Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση να το συζητήσω το θέμα, αλλά να ξέρουμε γιατί πράγμα συζητάμε και είναι κάτι το οποίο θα πάρει αρκετό χρόνο να οικοδομηθεί, να διοργανωθεί, ενώ το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα είναι άμεσο και πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα εμεί ω Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο να συνεργαστούμε με οποιοδήποτε περιφερειακό νομισματικό, ε, θεσμικό ίδρυμα όπω το Ευρωπαϊκό ε, Ενδυνάμει ε, ε, νομισματικό ταμείο. Είναι εδώ ε, μια προοπτική εφικτή να συνεργαστούμε με ένα περιφερειακό νομισματικό ταμείο σαν αυτό όταν θα αρχίσει να υφίσταται όπως ε, έχουμε και το θέμα της αντιμετώπισης κονδυλίων που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που διατίθενται για παράδειγμα σε άλλες χώρες όπως τη Λετωνία εκτός δηλαδή Ευρω... ζώνης ευρώ. Τώρα για το θέμα το οποίο έχουμε εδώ μπροστά μας σε σχέση με τις... Ε, αν μπορούσατε να απαντήσετε στα γαλλικά. Εντάξει, ευχαρίστω, θα το κάνω. Είναι περίπλοκο το θέμα. Είναι περίπλοκο να διαπιστώσουμε τα βαθύτερα αίτια της κρίσης. Τα άμεσα αίτια ήταν βεβαίως ε, το πρόβλημα με την αγορά κατοικίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και τα Βεβαίως, ένα ερώτημα είναι γιατί έχουν τόσα χρέη τα αμερικάνικα νοικοκυριά. Έχει να κάνει με τις ανισότητες ε, εισοδήματος, ε, έχει να κάνει με τις αυξήσεις των μισθών που είναι μικρότερες για τους πιο φτωχούς. Τώρα, το ενδιαφέρον είναι το τι συμβαίνει τώρα. Αυτή τη στιγμή η μεγάλη αλλαγή είναι η αποταμίευση των Αμερικανικών νοικοκυριών που γίνεται για πρώτη φορά. Σήμερα έχουμε περίπου 6-7% και ενδεχομένως να αυξηθεί στο 9-10% λένε κάποιοι άλλοι. Ακόμη όμως και αν παραμείνει για πολύ καιρό στο 6-7%, όχι για 6 μήνες, αν δηλαδή πρόκειται για μακροπρόθεσμη αλλαγή, μιλάμε για θεμελιώδη αλλαγή που θα έχει σημαντικές συνέπειες στις πιστώσεις, αλλά και σε αυτήν την περιβόητη ανισότητα ανισορροπία γιατί θα μειώσει το, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου και θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ισορροπία το σύστημα. Άρα αυτό είναι η... Η ανισότητα στους μισθούς είναι η ρίζα η βαθύτερη πολλών προβλημάτων. Όμως από εκεί και πέρα προκύπτουν και πολλά άλλα θέματα. Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο και το ΔΕΛΤΑ νομίζω ότι έχω απαντήσει γενικά. Τώρα, για τον φίλο τον κύριο Γκέμπελς στο θέμα της Βασιλείας. Εγώ νομίζω ότι έχει γίνει μέχρι στιγμή ήταν πολύ ποιοτικό. Και η εγγύηση είναι ότι συμμετέχει και το Νιτάφ. Το πρόβλημα όμως είναι ότι παίρνει χρόνο. Ας μην ξεγελιόμαστε. Θα πάρει χρόνο. Και ο αγώνας συνεχίζεται. Παραμένει λοιπόν αυτή η μεγάλη αντίφαση. Επιπλέον ελπίζουμε να έχουμε τελικά ένα παγκόσμιο σύστημα. Λογικά αυτό χρειάζεται, βεβαίως στην πράξη είναι συζητήσιμο το θέμα. Και να μην ξεχνάμε ότι η Βασιλεία 2 δεν εφαρμόστηκε από τους Αμερικανούς και ούτε και τώρα υπάρχει τέτοια τάση. Και αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα για τους υπόλοιπους. Εγώ θεωρώ ότι το προϊόν αυτής της κρίσης ήταν μια καλύτερη συνεργασία των διαφόρων κυβερνήσεων. Όμως, μην είμαστε αφελείς και να πιστεύουμε ότι τα εθνικά ή περιφερειακά συμφέροντα έχουν εξαφανιστεί. Ευχαριστώ αντιμετωπίζουμε μεγάλες δυσκολίες γιατί δεν νομίζω ότι θα έχουμε χρόνο να απαντηθούν οι ερωτήσεις που θα ακούσουμε. Θα προσπαθήσουμε όμως να τα καταφέρουμε. Ο κύριος Τζορτζέτη από την Ιταλία έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Τάχιστα ένα ερώτημα. Θέλω να αναφερθώ λίγο στην πραγματική οικονομία και διότι πιστεύω ότι σαν σταθερότητα του συστήματος κατά κάποιο τρόπο ε, φταίνε και και οι προϋπολογισμοί των χρησιμοποιητικών ιδρυμάτων. Θα ήθελα εξηγήσεις πώς από τη Βασιλεία 2 στη Βασιλεία 3 θα γίνει το πέρασμα. Το πρόβλημα των μικρομεσών επιχειρήσεων πώς λαμβάνεται υπόψη. Αν δεχτούμε ότι θα γίνει η πιο καλή δυνατή ανάκαμψη, κάτι που ευχόμαστε, χρειάζεται μεγαλύτερη. Πώ υπάρχει δυνατότητα να δίνουν περισσότερε πιστώσει οι τράπεζε, όσον αφορά σε σχέση πάντα με τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, είναι το ερώτημα. Ο κύριο Πιτέλα. Πρόεδρε, θα είμαι συντομότατος. Ένα ερώτημα προς τον κύριο Ντράγκε. Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική έναντι των κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ασχολείται τώρα με τη ρύθμιση των hedge funds. Αυτό είναι κάτι που ακυρώθηκε από το, τη διάταξη του ECOFIN το θέμα. Πώς θα γίνει η παρέμβαση στον τομέα και πώς θα μπορέσουμε να αντιταχθούμε ε, στις κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Και τι γίνεται με τα ΣΦΟΠ σε σχέση με τα κρατικά ομόλογα και όσον αφορά τη διαμάχη μεταξύ Βερολίνου και Παρισίων, όσον αφορά το που θεωρείται το γερμανικό οικονομικό μοντέλο και που θέτει σε κίνδυνο όλη την Ευρωζώνη λόγω των εμπορικών πλεονασμάτων. Ε, πιστεύετε ότι είναι δυνατό να υπάρξει συνεργασία, μια προσέγγιση οικονομική, ε, ισολογισμό των προπολογισμών και κατά πόσο θα καταβληθούν δέουσες προσπάθειες ούτως ώστε να υπάρξει μια κοινή ευρωπαϊκή οικονομική ανάπτυξη. Thank you very much. Uh, uh, Mr. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκέρχαρντ Σεκ από τη Γερμανία είναι επόμενος. Ευχαριστώ. Τρεις σύντομες ερωτήσεις. Κύριε Ντράγκη, κάνατε λόγο για μεταβατικές προθεσμίες που πρέπει να είναι αρκετά διακόπτει ο μιλητής. Θα ήθελα να επανέλθω σε κάποια σχόλια όσον αφορά τον Μάριο Ντράγκη, ώστε να μην χρειάζεται μετάφραση. Τώρα όμως φόρεσαν τα ακουστικά τους, Οπότε, εντάξει, τώρα στα γερμανικά και πάλι. <laughs> Θα ήθελα να αναφερθώ στην παρατήρηση του κυρίου Ντράγκη για τις κεφαλαιακές ανάγκες. Ε, προϋποθέσεις. Είπατε ότι πρέπει να είναι αρκετά μεγάλες οι Μου θυμίσει αυτό τη μοίρα των γερμανικών περιφερειακών τραπεζών που χρησιμοποίησαν την μεταβατική περίοδο ώστε δισεκατομμύρια ε, επικίνδυνων αξιών και χρεογράφων και ομολόγων να αγοράσουν. Ερώτηση, υπάρχουν κάποιοι κανόνες που έχουν συζητηθεί και εξεταστεί ώστε να αποφύγουμε ώστε αυτή η μεταβατική περίοδος να οδηγήσει σε νέα προβλήματα ώστε να μην οδηγήσει σε νέα προβλήματα αυτή η μεταβατική περίοδος. Η δεύτερη ερώτηση αφορά την σύνθεση αυτού του Global Risk Board Global Risk Στην Ευρώπη σχεδιάζεται να αποσταλούν ε, πολλοί εκπρόσωποι από τις Ευρωπαϊκές Κεντρικές Τράπεζες εδώ μια και δεν ήταν ιδιαίτερα σε γρήγορση η, Ευρω... η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα σε σχέση με την κρίση στέγασης, ποια είναι η στάθμιση των πραγμάτων, πώς πρέπει, ποια πρέπει να είναι η αναλογία των εκπροσώπων των κεντρικών τραπεζών σε ένα τέτοιο Global Risk Board. Τρίτη μου ερώτηση αφορά τον κύριο Στροσκάν. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον έγγραφο από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που αφορά το θέμα του πολιτικού lobbying και συζητά, εξετάζει αυτό το θέμα και λέει ότι το πολιτικό lobbying πρέπει να εξετάζεται ως ένα ε, ένας παράγοντας συστημικών κινδύνων. Πολύ ενδιαφέρον αυτό σε σχέση με αυτά που συνέβησαν στην κρίση στις ΗΠΑ. Υπάρχουν πολιτικά συμπεράσματα σε σχέση με αυτό από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πώς θα έπρεπε να αντιδράσετε σε ένα τέτοιο πόρισμα. Και αν μου επιτρέπετε μια τελευταία ερώτηση παρακαλώ πιστεύω πρέπει και πάλι να ξαναδούμε πώς δεδομένα, δεδομένων των ε, ολοκληρωμένων παγκοσμιοποιημένων αγορών θα αντιδράσουμε σε παγκοσμιοποιημένα θεσμικά όργανα και πώς ε, το κράτος υποδοχής θα μπορεί ίσως να ενισχύεται. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε κινδύνους από μια θηγατρική εφόσον η μητρική εταιρεία σε μια άλλη ήπειρο θα μπορούσε αυτή τη φερεγγιότητα, τη ρευστότητα από τη θηγατρική να την αφαιρέσει να την αποσύρει. Πώς μπορούμε εδώ να διασφαλίσουμε ότι ο εκπρόσωπος ε, της χώρας υποδοχής θα έχει αρκετές εξουσίες. Ευχαριστώ. Στόγιαν παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έχω μια πολύ σύντομη ερώτηση για τον κύριο Μάριο Ντράγκη Προφανές είναι ότι το χρηματοοικονομικό σύστημα σταθεροποιήθηκε χάρη σε μια τεράστια σταθεροποιητική προσπάθεια που απέτησε τεράστιον όγκο κονδυλίων. Τώρα διαπιστώνουμε ότι μια ολόκληρη σειρά δράσεων είχε γίνει σε σχέση με τοξικά ομόλογα και που συνεχίζονται. Παράδειγμα, επενδυτές που δεν έχουν κανένα τίτλο όσον αφορά ε, δάνεια, για παράδειγμα ε, όσον αφορά την Ελλάδα και που θεωρούν αναγκαίο να διασφαλιστούν σε σχέση με τους κινδύνους που απορρέουν από μια τέτοια χώρα. Ερωτώ, δεν πρέπει να σταματήσουν τέτοιες κερδοσκοπικές δράσεις με κάθε ταχύτητα, γοργότατα, διότι η αρχιτεκτονική του συστήματος ε, εδώ και αρκετό χρόνο ακολουθεί τέτοιες τάσεις και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ερώτηση προς τον κύριο Στροσκάν Κατανοώ ότι είσαστε σύμφωνος με την δημιουργία ενός ταμείου με κονδύλια, ενός νομισματικού ιδρύματος για παράδειγμα μελλοντικά για την εξυγίανση του τομέα των τραπεζών και ότι το τέλος στις τραπεζικές συναλλαγές που θα επιβάρυνε τις συναλλαγές θα μπορούσε να είναι μια πηγή άντλησης κονδυλίων για αυτό το ταμείο. Και τώρα ένα σχόλιο, ένα σχόλιο για αυτά τα οποία είπατε σε σχέση με τον πληθωρισμό προηγούμενα. Εγώ ε, έζησα μια περίοδο κατά την οποία το Λίμπορ έφτασε στο 17% με την κρίση την πετρελαιακή κατά την δεκαετία του 80 έναντι της πρόσφατης ε, κατάστασης. Η ερώτηση που θέλω να σας θέσω είναι το η εξής. Σε σχέση με εκείνες τις χώρες που συσσόρευσαν πάρα πολλά μεγάλα χρέη σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα όσον αφορά την αύξηση του χρέους τους, δεν θα έπρεπε να, τους προειδοποιήσουμε, να προειδοποιήσουμε αυτά τα κράτη και κάτι να κάνουμε. Ευχαριστώ. Ο κ. Σκινάρη από τη Φιλανδία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Στην Φιλανδία τη δεκαετία του 90 είχαμε μια πολύ άσχημη τραπεζική κρίση και μάθαμε κάποια πράγματα από αυτήν. Και γι' αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω η αισιοδοξία σας για το ότι ξεπεράσαμε αυτή την κρίση και ότι βγήκαμε αρκετά καλά από την κρίση. Σε τι βασίζεται αυτή η αισιοδοξία σας. Βλέποντας την κατάσταση των ευρωπαϊκών χωρών βλέπουμε ότι πολλές χώρες είναι στην χειρότερη κατάσταση που πέρασαν ποτέ από τη στιγμή που μπήκαν στο ευρώ. Και ταυτόχρονα στην Κίνα και στην Ινδία εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι ήρθαν από την Ήπεθρο και πήγαν στις πόλεις και εξακολουθούν να εργάζονται στις πόλεις και κάνουν τις ίδιες δουλειές που έκαναν παλιά στην Ευρώπη και στις Ηνωμένε Πολιτείες οι εισαγωγές μειώθηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, οπότε στην πράξη πώς θα προχωρήσουμε. Ταυτόχρονα το εποπτικό σύστημα στο οποίο αναφερόσασταν, αν σκεφτούμε την Ουάσιγκτον, όπου είναι η έδρα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και όπου συναντώνται κάθε μέρα αυτοί οι σημαντικοί άνθρωποι, συναντάτε αυτούς τους σημαντικούς ανθρώπους και το κάνατε και τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, θα πρέπει να μην ε, κοροϊδεύονται τα κράτη. Πώς θα αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα, να μην ξεφύγει η κατάσταση από τον έλεγχο σε κάθε χώρα. Και όσον αφορά, εφόσον αυξήθηκαν τα αποθεματικά, ε, πού βρίσκονται αυτά τα χρήματα όταν περιμένουμε την αύξηση των ε, επιτοκίων. Ποιος θα ωφεληθεί από αυτό, πιθανότατα όχι τα κράτη, τα εθνικά κράτη. Όσον αφορά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, άλλο ένα ερώτημα. Αν μια ευρωπαϊκή χώρα βοηθηθεί, πώς θα επηρεάσει αυτός, αυτό την ισοτιμία του ευρώ. Ευχαριστώ. Η Σιλβί Γκουλάρ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μία ερώτηση και για τους δύο και καταρχάς να σας ευχαριστήσω που παραμείνατε μαζί μας και περνάω στα γαλλικά ως εισηγήτρια για τους συστημικούς κινδύνους έχω μία απλή ερώτηση. Για το πακέτο του ελέγχου μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτό που τονίσατε. Μία Ευρώπη σε παγκόσμιο επίπεδο. Εμείς διαπιστώνουμε τρεις αλλαγές καταρχάς ο πρόεδρος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας να είναι στην Προεδρία του Ταμείου. Δεύτερον, μεγαλύτερη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και τρίτον, στην Φραγκφούρτη να εξετάζονται όλοι οι δείκτες μικροοικονομική και μακροοικονομική της ευρωπαϊκής οικονομίας. Θεωρείτε ότι αυτές οι προτάσεις είναι επαρκείς ή έχετε να προτείνετε και κάτι άλλο που θα μπορούσαμε να προτείνουμε εμείς ως εισηγητές του Κοινοβουλίου. Κύριε Μπερές, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους δύο μιλητές. Τρεις ερωτήσεις. Καταρχάς, βλέπουμε τις ε, μεταρρυθμίσεις ε, στις ε, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες μετά την κρίση και βλέπουμε ότι ο δημόσιος τομέας βοήθησε τον τραπεζικό τομέα και υπήρξε μεγάλη αναστότωση. Έχουμε τώρα το πακέτο για τον έλεγχο όμως, συμφωνώ με τον κύριο Τράγκη ότι υπάρχει ο κίνδυνος όλοι να προτείνουν τη δική τους ε, ιδέα και τελικά να κάνουμε ένα μείγμα που δεν θα βοηθάει κανέναν. Από τη μία πλευρά λέμε να συγκεντρωθούν όλες οι ήπειροι και να καταλάβουν και οι πολίτες ότι υπάρχουν ε, κίνδυνοι που σημαίνουν ότι χρειάζεται αλληλεγγύη για να καταφέρουμε ε, κάτι. Όμως ένα θέμα είναι η φορολογία των τραπεζικών χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Αλλά πού θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα ρωτάνε. Τι μας ενδιαφέρει αυτό. Υπάρχει εδώ μια δημόσια συζήτηση επί της οποίας πρέπει να προχωρήσουμε. Και θέλουμε να μπορέσουν τελικά οι Υπουργοί να καταλήξουν σε μια χρήσιμη πρόταση γιατί είναι θέμα ευθύνης μας απέναντι στους πολίτες χωρίς να χρειαστεί να περιμένουμε το τι θα γίνει με το πακέτο που έχουμε αυτή τη στιγμή επιτάπητος. Όσον αφορά τα CDS, άκουσα την απάντηση του κυρίου Ντράγκη και δεν μπορώ να συμφωνήσω με την ιδέα ότι όλα τα CDS πρέπει να βρίσκονται σε... στις ΙΠΑ, να ρυθμίζονται από τις ΙΠΑ. Το αποτέλεσμα από κάτι τέτοιο είναι ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να ζητήσει διαφάνεια, να γνωρίζει ακριβώς τι συμβαίνει και στην πράξη. Άρα τα πράγματα είναι πολύπλοκα και νομιμοποιείται η Ευρώπη να ζητάει περισσότερα όσον αφορά τη σύνθεση μιας ελεγκτικής αρχής των CDS. Και ένα άλλο θέμα όσον αφορά το δημοκρατικό διάλογο. Νομίζω ότι όλοι έχουμε καταλάβει από τις συζητήσεις ότι υπήρχαν πολλές συγκρούσεις συμφερόντων και από αυτές προέκυψε αυτή η απορρίθμιση. Όμως, εγώ βλέπω έναν κίνδυνο να αποκλειστούμε εμείς από τις συζητήσεις. Πού είναι ο δημοκρατικός διάλογος. Πού θα μπουν τα στοιχεία για τον επαναπροσανατολισμό των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Εμείς θέλουμε ένα τομέα ο οποίος θα μπορεί να επιτρέψει και την ανάπτυξη και να λάβει υπόψη και τη γύρανση του πληθυσμού. Πού θα γίνει η συζήτηση, γιατί πρέπει και εμείς να συμμετέχουμε και να δώσουμε απαντήσεις, αλλά βεβαίως θέλουμε να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις. Ευχαριστώ κύριε Καλμάρη, Φιλανδία. Ευχαριστώ έλαβα απαντήσεις σε ερωτήσεις που ήθελα να αποβάλω. Θα ήθελα απλώς να σε ενθαρρύνω να δημιουργήσετε διεθνή φόρο των συναλλαγών των διεθνών χρηματοστοτικών αγορών για την αντιμετώπιση των κινδύνων. Δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουν, να υπομίζονται τον κίνδυνο τα κράτη-μέλη στον αφορά τους κινδύνους. Ευχαριστώ και φτάνω με την Άντελίν Σάντσες Πρεσέδο. Ευχαριστώ πολύ. Προς τον κύριο Τράγκη, παρότι όλοι οι φορείς σε κάποιους όρους μπορούν να δημιουργήσουν συστημικούς κινδύνους, μπορούν να υπάρχουν κάποια χρηματοοικονομικά θεσμικά όργανα που μπορούν να προκαλέσουν συστημικούς κινδύνους παγκόσμια. Θα πρέπει να ταυτοποιηθεί πολυμερώς αυτό. Μπορεί να γίνει. Δεύτερον, για τις ε, υπηρεσίες για ε, τους ε, αξιολόγησης σε σχέση με την αμεροληψία οι υπηρεσίες αυτές αξιολόγηση αξιολόγησης εντάσσονται στην αγορά και αντανακλούν και συμφέροντα σε σχέση με την αγορά. Αυτό δεν είναι ασύμβατο σε σχέση με την αξιολόγηση δημοσίων φορέων. Η, και για κάποιες ανισορροπίες που υπάρχουν. Μου φάνηκε ότι είσαστε πολύ αισιόδοξο σε σχέση με το πολυμερές πλαίσιο ότι αυτά τα οποία συνέβησαν σε σχέση με το εμπόριο μπορούν να επιτευχθούν και σε σχέση με το χρηματοοικονομικό τομέα. Ερώτηση, στους, στο νομισματικό τομέα μιλήσαμε εδώ για την, τις ανισότητες ε, σε σχέση με τις διάφορες χώρες. Πώς μπορούν τα, οι ανισότητες αυτές ε, να εξισορροπηθούν ε, με ένα τρόπο καινοτόμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτός ήταν ο τελευταίος γύρος ερωτήσεων και μας έμειναν και κάποια θέματα από τον προηγούμενο γύρο. Σχόλιο για το μέγεθος των τραπεζών σε σχέση με τη χώρα. Δεν είμαι σίγουρη αν απαντήθηκε αυτό. Κύριε Τρασκάν, μήπως να ξεκινήσετε τις απαντήσεις. Ναι, ευχαριστώ. θα υπάρχουν και ερωτήσεις που αφορούν τα CDS και ίσως ο Μάριο θα πρέπει να απαντήσει περισσότερο ως αυτό το θέμα. Το θέμα αυτό των πολιτικών, του πολιτικού lobbying πάντα υπήρχε σύγκρουση με το, μεταξύ των διαφόρων κοινοβουλίων των διαφόρων κρατών μελών για το ποιο είναι ο νόμο από τη μία πλευρά και των ιδιωτικών συμφερόντων προσπαθούν να επηρεάσουν τα τεκτενόμενα. Δεν βλέπω να υπάρχει στην πράξη μεγάλο πρόβλημα. Αυτό είναι κανονικό. Οι κοινοβουλευτικοί να έχουν τι καλύτερε πληροφορίε και οι καλύτερε πληροφορίε προέρχονται από αυτού που άμεσα εμπλέκονται στι επιχειρήσει. Διαφορετικέ πληροφορίε, σύγκρουση πληροφοριών κλπ. Το πρόβλημα πού έγκυται. Αν τυχαίνει αυτό που θες να κάνεις σε πολιτικό επίπεδο δεν μπορεί να γίνει λόγω πολύ μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων. Και αυτό είναι ένα ερώτημα που ξεπερνά τα όρια της αναδιάθρωσης χρηματοδοτικού τομέα. Μπορεί το ίδιο να τίθεται σε διάφορους άλλους τομείς. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Διότι αυτή την περίοδο όλοι αναφερόμαστε στο συστημικό κίνδυνο και θα ήταν ενδιαφέρον να εξετάσουμε και άλλους συστημικούς κινδύνους εκτός από τους παραδοσιακούς που προέρχονται από το τραπεζικό τομέα. Όσον αφορά τις υποπτικές αρχές των χωρών υπάρχει πρόβλημα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ε, ασχολείται με τη διασυνοριακή επίλυση και το πρόβλημα που είχα αυτή την κρίση που τοποθετούτο. Εάν είχαμε διασυνοριακή επίλυση προβλημάτων πολλές μητρικές ε, χώρες είχαν θηγατρικές σε πολλές χώρες, ε, είχαν θηγατρικές σε Και είναι κατανοητό ότι αν έχουν πρόβλημα στην βάση, επιλύουν το πρόβλημα στη χώρα, αλλά δημιουργούνται προβλήματα εκεί που είναι οι θηγατρικές. Ποιος ρυθμίζει το όλο θέμα είναι το πραγματικό πρόβλημα. Και η εποπτική αρχή μιας χώρας ίσως να μην δίνει λύση σε όλα τα προβλήματα Διστάζω. Δεν θα ήθελα να έχω ένα σύστημα που βασίζεται σε αυτή την ιδέα. Και υπάρχει και κάτι άλλο που μπορούμε να πούμε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Σε αυτή την κρίση. Μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία ανελήφθη. Η πρωτοβουλία της Βιέννης, όπως αποκαλείται μέχρι ότου να την αναλάβει περισσότερο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποια ήταν η ιδέα, να συναθιστούν ιδιωτικέ τράπεζε, το Διεθνέ Ταμείο, κεντρικέ τράπεζε, το FSB και όλοι μαζί να πούμε ότι, ότι εάν έχετε επενδύσει όλε τι δυτικέ τράπεζε στην Ανατολική Ευρώπη και πάρετε τα χρήματά σα, θα καταρρεύσουν αυτέ οι χώρε. Σαν τράπεζε μπορεί να πείτε αυτό δεν είναι δικό μα πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα, ότι αν υπάρξει αυτή η κατάρρευση στην κεντρική Ευρώπη, θα έχει αντίκτυπο επάνω σα. Άρα τελικά καταστρέφει τον εαυτό σα. Και λειτουργεί αυτό, αλλά δεν, όχι 100%, αλλά λειτουργεί αυτή η προσέγγιση. Το τραπεζικό σύστημα κατάλαβε, ο τραπεζικό τομέα κατάλαβε ότι θα πρέπει να κρατήσουν τι ροέ του στι χώρε που έχουν πρόβλημα στην κεντρική Ευρώπη, διότι ήταν κομμάτι του γενικού προβλήματο και αν υπάρχει το πρόβλημα εκεί ίσω να επηρεάσει την υπόλοιπη Ευρώπη. Το θέμα δεν είναι μόνο ποιο είναι επόπτη, αλλά θα πρέπει να υπάρξει θεσμός που δημιουργεί λύσεις διασυνοριακές και να μην ξεχυλίζουν τα προβλήματα από μια χώρα και να επηρεάζουν τις γύρω χώρες. Είναι κάτι που επεξεργαζόμαστε αλλά δεν έχει επιλύθει ακόμα το πρόβλημα. Τώρα το άλλο ερώτημα, ερωτήματα που ετέθησαν από διάφορες πλευρές για το FTG, τον φόρο για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Εγώ ήμουν υπέρμαχος αυτού του φόρου τη δεκαετία του 70. Έκτοτε πολλά άλλαξαν. Και συγκεκριμένα αυτό που άλλαξε είναι αυτό που συζητούμε σήμερα το πρωί, αυτό που κουβεντιάζουμε ήδη τις ώρες. Δηλαδή τεχνικές λεπτομέρειες που διέπουν ε, το χρηματοστητικό τομέα. Και το επεξεργαζόμαστε, ακολουθώντας εντολή που μας δόθηκε από τους G20, όπως είπε η κυρία Περέζ. Εξετάζουμε κάθε φόρο του χρηματοστητικού τομέα συμπεριλαμβανομένων των χρηματοστατικών συναλλαγών, αλλά και άλλου φόρου και συναλλαγέ, να δουν ποια είναι τα υπέρ, ποια είναι τα κατά. Αυτό είναι προφανέ και δεν μπορώ να σα δώσω συμπέρασμα τώρα. Το συμπέρασμα θα το έχουμε σε 1,5 μήνα. Αλλά αυτό που διαφαίνεται είναι το εξή. Γίνεται όλο και πιο εύκολο να δημιουργούνται οι παράγωγα για να αποφευθεί ο φόρος των συναλλαγών και τέλος το ελκυστικό αυτού του φόρου μπορεί να αντισταθμίζεται από το ότι δεν θέλει κανείς να δημιουργήσει ένα φόρο και ένα σύστημα που στο τέλος θα το αποφεύγουν οι περισσότεροι φορείς διότι μπορούν να βρουν έναν τρόπο να ξεφύγουν. Όσον αφορά τη φορολόγηση, όσο πιο απλά είναι τα πράγματα, τόσο το καλύτερο. Το απλούστερο είναι το καλύτερο. Και αν θες να κάνεις κάτι, αν είναι πολύ γερό, άκομψο ίσω θέμα είναι πιο εύκολο να εφαρμοστεί και αν είναι πολύ λεπτομερές, πολύ προωθημένο, έχει πολλά κενά. Δεν καταλήγω σε συμπέρασμα τώρα. Αλλά δεν είναι και τόσο προφανές ότι η μοναδική λύση περνάει από ένα φόρο συναλλαγών. Υπάρχουν υπέρ και κατά, αλλά ίσως να είναι ευκολότερο. Ο στόχος είναι να μειώσουμε την επικίνδυνη συμπεριφορά στο χρηματοστηρικό τομέα, να εισαγάγουμε περισσότερα διοντολογικά στοιχεία στον τομέα ή να παράγουμε πόρου που μπορεί να χρησιμοποιηθούν όπω θέλει κάποιο. Γι' αυτό που έχει προτεραιότητα δεν είναι τόσο προφανέ ότι το ευκολότερο είναι να δημιουργήσουμε κάτι που ίσω και είμαι προσεκτικό θα το λέω, που ίσω λέω να είναι δύσκολο να δημιουργηθεί και αρκετά εύκολο να υπερκεραστεί, να αποφευχθεί. Άρα εκρεμεί το θέμα στο έγγραφό μας και το έγγραφό μας θα είναι έτοιμο τον Απρίλιο. Σίγουρα θα δώσουμε απαντήσεις. Θα πούμε ότι υπάρχει περιθώριο για κάποιο φόρο του χρηματοπιστωτικού τομέα, δεν ξέρουμε όμως τι φόρο θα προτείνουμε. Ίσως εδώ να διαφωνώ εδώ με τον συνάδελφο, η εξισορρόπηση μεταξύ ρύθμισης και φορολόγησης. Ποια είναι. Κάποιοι, πολλοί μάλλον, οι κεντρικές τράπεζες, οι διευθυντές των κεντρικών τραπεζών λένε ότι μπορεί να κάνεις τόσα πολλά με ρύθμιση που δεν χρειάζεται φορολόγηση. Είναι ένα επιχείρημα που μπορεί να ληφθεί υπόψη. Είναι σωστή ισορροπία. Τι προέρχεται από ρύθμιση. Ρύθμιση τενό, Εποπτεία, ρύθμιση, έλεγχο κλπ. Και όλα αυτά και απ' την άλλη αυτά που προέρχονται από ένα φορολογικό σύστημα που είναι πιο υποχρεωτικό, πιο περιοριστικό σύστημα, αυτά τα δύο πρέπει να εξισορροπηθούν, πρέπει να συζητηθεί αυτή η ισορροπία. Άλλο ερώτημα που αφορούσε αποτελεσματική χρηματοστική αγορά στην Ευρώπη για το μέλλον. Αυτό χρειάζεται όχι μόνο η Ευρώπη, αλλά σίγουρα η Ευρώπη. Έχει τεράστιες επενδύσεις περιμένει τεράστιες επενδύσεις και εφαρμογή του προγράμματος της Λισαβόνας αγαλλικά. Το ξέρω ότι θα έχω πρόβλημα. Καλώς. Ας αλλάξω. Ας μιλήσω γαλλικά τώρα. Ίσως και μη γαλλόφωνοι θα καταλάβουν καλύτερα τα γαλλικά μου από τα αγγλικά μου. Προφανώ η Ευρώπη χρειάζεται πιο αποτελεσματική χρηματοστική αγορά και έχει μπροστά τη χρηματοδοτήσεις κολοσιέ και προς τις δύο κατευθύνσει που ανέφερε η Περβάνς. Καινοτομία, ανταγωνιστικότητα και για να προχωρήσουμε για εκάλυψη του προβλήματος της γύρανση του πληθυσμού από την άλλη. Όμως το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε πάντα να έχουμε στόχους αντιφατικούς. Αν θέλουμε χρηματοστικές αγορές που είναι αποτελεσματικές, δεν θα πρέπει να χρονοτριβούμε λέγοντας ότι οι αγορές αυτές είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Θα πρέπει να καταλήξουμε σε χρηματοστικές αγορές ρυθμισμένες, χρηματοστητικές αγορές που δεν ξεφεύγουν από αυτά που δημιουργήσαμε, που δεν παράγουν συνέπειες αντίθετες από αυτές που θέλουμε, αλλά κάνοντας αυτά να μην σκοτώνουμε κιόλα τις αγορές εκείνες που επιτρέπουν τις επενδύσεις. Διότι το πραγματικό πρόβλημα είναι να έχουμε σωστή κατανομή των αποταμιεύσεων. Λοιπόν, για να μην χρονοτριβώ, δεν θα μου αφήσει χρόνο η Πρόεδρος, δεν είμαι πραγματικά πεπισμένος ότι η, η, κατανο, η ε, είναι αποτελεσματική η χορήγηση, η, το μετάβαση από τι αποταμίες ευρωπαϊκές προς επενδύσεις. Χρειαζόμαστε λοιπόν στην Ευρώπη δημιουργία ενός συστήματος χρηματοδότησης που να είναι διαφορετικό, αποτελεσματικότερο από αυτό που έχουμε σήμερα. Υπάρχουν πάντα αντιφάσεις, αντιθέσεις, να κάνουμε αυτό και ταυτόχρονα θέλουμε να πλαισιώσουμε καλύτερα τις χρηματοστηρικές αγορές για να αποφύγουμε παρεκκλήσεις κλπ. Αυτό είναι πάρα πολύ περίπλοκο και δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε κανένα του δύο πυλώνε. Κανένα δεν θέλει να εγκαταλείψει κανεί την ιδέα ότι χρειάζεται καλύτερη ρύθμιση των αγορών, αλλά κανεί Επίσης δεν θέλει να πει ότι ε, θα αφήσουμε ελεύθερες στις ε, χρηματιστικές αγορές και θα βρούμε άλλες μορφές για να περνάνε οι αποταμιεύσεις στις επενδύσεις χωρίς να χρειαζόμαστε τις χρηματιστικές αγορές. Είναι καλό ότι αυτή η άποψη έχει εξαφανιστεί. Πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ των θέσεων. Αυτή η ισορροπία έχει και το κόστος της. Αυτή η ισορροπία δεν περνά υποχρεωτικά από τους ίδιους μηχανισμούς στα διάφορα μέρη του κόσμου. Μπορεί να υπάρχουν διαδικασίες κατανομής λειτουργίες αγοράς που δεν είναι διαφορετικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ιαπωνία κλπ. Γι' αυτό, για το κόστος, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια είναι πάρα πολύ σημαντικός. Διότι υπάρχουν πράγματα που διευθετούνται καλύτερα, θέματα επικουρικότητας που ρυθμίζονται καλύτερα σε περιφερειακό επίπεδο από ό,τι σε παγκόσμιο επίπεδο τελευταία λέξη, το πρόβλημα του πληθωρισμού και τις υπερχρεωμένες χώρες. Είναι πάντα... Α, θα επιστρέψω στα Είναι πάντα πειρασμός για χώρες να επιλύουν τα προβλήματα δημοσίου χρέους με μεγάλο πληθωρισμό. Ποιο είναι το μειονέκτημα του μεγάλου πληθωρισμού. Ότι δεν πετυχαίνει σωστά ωφέλη, αρκετά ωφέλη μέσω αυτής της μεθόδου. Για τα μεγάλα χρέη, δημόσια χρέη, που οι περισσότερες χώρες στην Ευρώπη αντιμετωπίσουν τώρα, εγώ προτείνω να προσπαθήσουν να το λύσουν, να μην το λύσουν μέσω πληθωρισμού. Ένα παράδειγμα. Σύντομα θα μπορείτε να σα το στείλω με τα χαράς, αλλά θα το βρείτε και στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, θα βρείτε ένα πολύ ενδιαφέρον έγγραφο. Που τι δείχνει το έγγραφο. Έτσι γενικά, σε προχωρημένες οικονομίες, χρέος, ο λόγος χρέο ΑΕΠ θα έχει αυξηθεί το, 20, το 2014 σε, 4, σε 3 χρόνια σε 110% κατά μέσο όρο. 35% περισσότερο από ό,τι πριν από την κρίση. Και δεν είναι τύπο αμεληταίο το 35%. Αλλά το 10%, 35% είναι αυτό που δίνεται για την τόνωση της οικονομίας και τα υπόλοιπα είναι από την κρίση. Γιατί το λέω αυτό, διότι βλέπω να ακούγονται διάφορα σχόλια που λένε ότι το χρέος θα είναι τόσο ψηλό σε λίγα χρόνια διότι αυτό είναι συνέπειες των μέτρων ε, τόνωσης που ε, Αντίθετα, χωρίς την τόνωση αυτή θα ήταν βαθύτερη κρίση και με τη βαθύτερη κρίση θα είχαμε μεγαλύτερη χρέωση. Αυτό το συζητήσουμε τους επόμενους μήνες. Είναι κάτι ενδιαφέρον το οποίο ήθελα να υπογραμμίσω. Όλα τα άλλα ερωτήματα είναι για τον Μάριο να απαντηθούν. Μπορώ να πάω και μετά μπορώ να πάω σπίτι μου, λέει ο κύριος Μάριο. Ευχαριστώ. Πολλές ερωτήσεις αφορούσαν τα CDS. Συνοπτικά θα μπορούσα να απαντήσω ως εξής. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ε, τρεις λέξεις συνθήματα. Πρώτον, να γνωρίσουμε. Να γνωρίσουμε τι είδους αγορά είναι αυτή. Τα CDS και τα υπόλοιπα παράγωγα. Εκεί χρειαζόμαστε την στήριξή σας προκειμένου να αντισταθμίσουμε όλους αυτούς που έχουν συμφέροντα να αποφύγουν την κεντρική συναλλαγή το κεντρικό εμπόριο αυτών των παραγόγων. Όχι ότι αυτό είναι εύκολο, αλλά η κεντρική συναλλαγή σημαίνει μεγαλύτερη ορατότητα διαφάνεια, αλλά και για πολλές ε, τράπεζες σημαίνει απώλεια εσόδων. Και εκεί χρειάζομαστε τη στήριξη των κοινοβουλίων, των ομοθωτών. Το δεύτερο σύνθημα είναι απόφαση. Αν γνωρίζουμε μπορούμε να αποφασίσουμε ποια συμβόλαια θα είναι αποδεκτά και ποια όχι. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να απαγορεύσει κανείς κάτι το οποίο δεν γνωρίζει. Τότε μόνο θα αποφασίσουμε λοιπόν όχι μόνο ποια συμβόλαια θα είναι αποδεκτά, αλλά και ποιες απαιτήσει κεφαλαίου θα έχουμε για κάθε παράγωγο που θα εμπορεύεται. Γιατί ενδεχομένως δεν θα θέλετε να έχετε τις ίδιες απαιτήσει για όλα γιατί ορισμένα μπορεί να είναι πιο διαφανή και άρα να χρειάζονται διαφορετικές προϋποθέσεις. Και τέλος πρέπει να αποφασίσουμε ποιοι είναι οι αποδεκτοί αντισυμβαλόμενοι. Με ποιες προδιαγραφές θα πρέπει να συμμορφώνονται και ποιες θα πρέπει να είναι οι δεσμεύσεις τους. Και το τρίτο σύνθημα είναι ανταγωνισμός. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι θα ήταν χρήσιμο να έχει οργανισμό συμψηφισμού, ας το κάνει. Δεν ξεκινάμε από το μηδέν εδώ. Έχει γίνει ήδη πολλή δουλειά και δεν θα με εξέπλητε αν έβλεπα έναν ευρωπαϊκό οργανισμό συμφισμό και ενώ ευρωπαϊκό της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί ήδη υπάρχουν στην Ευρώπη οργανισμοί ψηφισμού στο Λονδίνο. Θα μπορούσε λοιπόν και θα ήταν καλό να υπάρξει τέτοιος οργανισμός συμψηφισμού. Όσον αφορά τα hedge fund, αυτό αφορά την περίμετρο της νομοθεσίας. Υπάρχει σκέψη για το πώς θα μπορούσαμε να επεκτείνουμε τις ρυθμίσεις και την νομοθεσία που ήδη υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες στα hedge fund. Και μπορώ να πω ότι υπάρχει σύγκληση αυτή τη στιγμή των νομοθεσιών. Έγινε πραγματική προσπάθεια το τελευταίο χρόνο για σύγκληση αυτών των νομοθεσιών. Οπότε είμαι αρκετά αισιόδοξο. Και να πω ότι η παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο FSB πραγματικά εμπλούτησε τον διάλογο και με τις υπόλοιπες αρχές, αμερικανικές, ιαπωνικές κτλ. και σε άλλους τομείς όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αν πρόκειται να έχουν διακριτική μεταχείριση όσον αφορά τις πιστώσεις από τη Βασιλεία 3, η απάντηση είναι όχι. Η Βασιλεία 3 θα επικεντρωθεί στις μεγάλες τράπεζες ε, και άλλες επιχειρήσεις ε, συναλλαγών. Και έτσι πρέπει να έχουν τα πράγματα γιατί όλοι μας είμαστε πεπισμένοι ότι η κρίση δεν ξεκίνησε από την παραδοσιακή διαδικασία πιστώσεων, αλλά κυρίως από τις κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, τα subprimes και τα Και εκεί επικεντρώνει τη Βασιλεία 3. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό θα δημιουργήσει κινδύνους για τις πιστώσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτή τη στιγμή θέλουμε να δημιουργήσουμε τράπεζες που θα είναι ανθεκτικές στις κρίσεις. Όπως είπε και ο Ντομινίκ, δεν ξέρουμε πότε θα έρθει η επόμενη κρίση, ούτε και από πού θα έρθει. Γι' αυτό πρέπει να δαπανίσουμε πολύ περισσότερη ενέργεια τώρα προκειμένου το σύστημα γενικά να είναι ανθεκτικό. Και επανέρχομαι στην κεντρικοποίηση των παραγόγων ως ένα παράδειγμα του τι μπορούμε να κάνουμε για να αυξήσουμε την ισχύ του συστήματος. Όσον αφορά τις απαιτήσει για την κεφαλαιοποίηση και τη μεταβατική περίοδο. Θα μπορούσαμε να δούμε τη διαδικασία της Βασιλείας 3 που συνεχίζεται με βάση το χρονοδιάγραμμα και άρα τώρα περνάμε στην εφαρμογή και η εφαρμογή από τις εθνικές αρχές πρέπει επίσης να γίνει με βάση το χρονοδιάγραμμα και να μην υπερβεί τα χρονοδιάγραμματα. Λοιπόν, η Βασιλεία 3 μπορούμε να πούμε ότι επικεντρώνεται σε δύο θέματα. Καταρχάς, επικεντρωνόμαστε σε ορισμένες παραμέτρους που αφορούν την κεφαλαιοποίηση, τη ρευστότητα και τις σχετικές απαιτήσει. Και αυτό από άποψη ορισμών δεν είναι περίπλοκο, αλλά είναι περίπλοκο από άποψη στάθμισης. Το άλλο θέμα όμως είναι η ποιότητα του κεφαλαίου, δηλαδή ποιες συνιστώσεις θα δημιουργήσουν τον ορισμό του κεφαλαίου, έναν ορισμό ο οποίος θα πρέπει να είναι παγκοσμίως αποδεκτός. Για πρώτη φορά δηλαδή θα πρέπει να έχουμε έναν ορισμό για το κεφάλαιο που θα είναι αποδεκτός παγκοσμίω. Βεβαίω όλοι ξεκινάμε από διαφορετικό σημείο εκκίνησης γιατί κάθε χώρα έχει διαφορετικό ορισμό. Εμείς καταλήξαμε σε μια συμφωνία, αλλά τι θα γίνει τώρα, σε μια νύχτα θα αλλάξουμε τον ορισμό του κεφαλαίου για όλους. Αυτό δεν γίνεται. Άρα πρέπει να δώσουμε χρόνο και στις τράπεζες και στις ελεγκτικές αρχές να προσαρμοστούν στο νέο ορισμό. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η μεταβατική περίοδος. Πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη ώστε οι τράπεζες να μην μπορούν να διαφορήσουν για μια αλλαγή που θα γίνει στο μέλλον. Και αυτό βεβαίως αποτελεί κομμάτι της συνολικής συμφωνίας. όσον αφορά τους, ε, τις ελεγκτικές αρχές ε, στην χώρα υποδοχής. Κοιτάξτε, το προηγούμενο χρόνο δημιουργήσαμε sovereign colleges, σώματα δηλαδή όπου συμμετέχουν οι ελεγκτικές αρχές ε, των κρατών. Και νομίζω ότι έχουν γενικά αν όχι επιλύσει το πρόβλημα τουλάχιστον ε, μειώσει σημαντικά το πρόβλημα. Να πω πάντως ότι αυτή τη στιγμή το σύστημα των μνημονίων αλληλοκατανόησης λειτουργεί αρκετά καλά προκειμένου να ρυθμίζει τα προβλήματα. Όσον αφορά τη συμμετοχή των κεντρικών τραπεζών στα risk boards, τα συμβούλια κινδύνων. Κοιτάξτε, οι κεντρικές τράπεζες ήταν από τις πρώτες που τόνισαν τη σημασία της κρίσης. Μπορείτε να δείτε τις δηλώσεις του 2004 και 2005 της ΕΚΤ και της ΕΦΑΙΕΣ όπου αναγνώριζαν και εντόπιζαν σιγά σιγά την κρίση. Υπάρχει λοιπόν τεχνογνωσία και εμπειρίες στην ε, Κεντρική Τράπεζα και γι' αυτό λοιπόν θα υπάρξει εκπροσώπηση και στην ECR, ESRB γιατί θα συμμετέχουν και οι τρεις προέδροι. Νομίζω ότι τελείωσα εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω τους ομιλητές μας που απάντησαν σε τόσες ερωτήσεις. Να ευχαριστήσω επίσης και τους ε, βουλευτές για την υπομονή τους. Δεν θα προχωρήσω σε σύνοψη γιατί χρησιμοποίησα το χρόνο για να ακούσουμε τους ομιλητές. Πάντως ζούμε σε ενδιαφέροντες καιρούς, πρέπει να εφαρμόσουμε πολλά και πρέπει να μάθουμε πολλά και να ανακαλύψουμε πολλά. Σας ευχαριστώ για την παρουσία, για την παρουσία σας και αναμένω με ανυπομονησία την επόμενή μας συνάντηση του χρόνου. <laughs>